Damen und Herren, ich darf die Sitzung eröffnen. Gibt es... Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Ξεκινάει η συνεδρίαση. Υπάρχει τίποτα για τη μερίσια διάταξη. Ναι, παρακαλώ κυρία Λούνατσεκ. Πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία, να ζητήσω συγγνώμη, ξέχασα την κάρτα μου στην Ολομέλεια. Οπότε παρακαλώ να μετρήσετε την ψήφο μου. Ε, είναι 8 η ώρα τώρα, τι θέτε. Νομίζω μπορείτε να πάτε στην Ολομέλεια να τη φέρετε και θα έχετε έρθει μόλις τελειώσει η ψηφοφορία. Και θα μετρήσουμε τη ψήφο μόνο εάν είναι σωστή. αλλά ξέρω και κάποιον άλλον που ψάξε την κάρτα του. Εγώ. We have Laila and Arif Yunis here today and yesterday in Strasbourg. Έχουμε τη Λαϊλά Γιουνίους εδώ πέρα, χθες και σήμερα, και ξέρετε πως ως Επιτροπή Εξωτερικών μας έχει απασχολήσει. Είχε προταθεί για το βραβείο Ζαχάροφ το 2014. μετά την ε, φύλαξή τους και καταφέραμε να βοηθήσουμε ιατρικά μέσω μιας ε, φιλανθρωπικής οργάνωσης ε, και της Κομισιόν και νομίζω ο Δόκτωρ Βίτ εκεί πέρα έκανε ό,τι μπορούσε για να σώσει ζωές και βεβαίως καλό είναι το ότι απελευθερώθηκε και ζει τώρα ζουν τώρα στην Ολλανδία όπου είναι οι κόρη τους ε, και έχουν λάβει άσυλο από τις Ολλανδικές αρχές. Επίσης, αυτό κατέστη δυνατό μετά από μακροσκελείς διαπραγματεύσεις με τις αρχές του Αζερβαϊτζάν. Μετά τη θεραπεία στο Βερολίνο τώρα έχουν βγει από το νοσοκομείο. Έχει ακόμα κάποια προβλήματα υγείας, αλλά νομίζω πως πρέπει να τους καλωσορίσουμε εδώ σε 9.45 στο τέλος της ε, συνεδρίασής μας για να τους ε, καλωσορίσουμε απλά για λίγα λεπτά και να τους ακούσουμε. Σας ευχαριστώ. Να τελειώσω, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα ταυτόχρονα Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για τη δουλειά που είχε, για τον συνάδελφο για τη δουλειά που είχε κάνει, γιατί χωρίς αυτόν δεν θα ήταν δυνατόν. Yes, chair. Κυρία Λούνατσεκ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς για τα όσα κάνατε έτσι ώστε η Λεϊλά και ο Αριφ να βγουν από τη φυλακή και να είναι σήμερα εδώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία. Σχέδιο γνωμοδότησης για την πρόταση κανονισμού και τα λοιπά, τα ξέρετε. Την έκθεση Βόλσκι. Έχετε να πείτε κάτι. Πριν από την εκτέλεση. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ψηφίσετε υπέρ ε, ε, μαζικά και με ενθουσιασμό γιατί το αξίζει η Ουκρανία. Ah, for the amendments. Oh, he's against Schafauer amendment. <laughs> Surprise. so, who is for the amendments 1 and 2. Τροπολογίες 1 και 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Η έκθεση στο σύνολό τη υπέρ ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Ναι, όχι, συγγνώμη, ενώ άρχεται. Πέρας. 42 υπέρ, 3 ε, ψήφοι κατά, 6 εποχές. Περνάμε τώρα. Τρίτες χώρες, οι υπήκοοι των οποίων πρέπει να έχουν θεωρήσεις. Έκθεση Μάμικινς. Γεωργία. Υπέρ των τροπολογιών 1 και 2. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την πρόταση. Άρχεται. Πέρας. 43 ε, υπέρ, 5 κατά, 3 αποχές. Συγχαρητήρια. Κοσφοπέδιο. Εδώ ο κύριος Επιτίδιος και ο Σαφάουερ θα έχουν στήριξη νομίζω. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το όλο πράγμα εκεί. Άρχεται η ψηφοφορία. καλησπέρας 38 υπέρ, 7 κατά 6 αποχές. Κυρία Λουνατσέκ, συγχαρητήρια, ζητήστε και το λόγο. Με ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ όλους που το στηρίξατε. Ζήτησα το λόγο γιατί, όπως ξέρετε, η Επιτροπή Αστικών Ελευθεριών, η Τάνια Φαγιών, ζήτησε να αναβληθεί η ψηφοφορία στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που είναι υπεύθυνη από την επόμενη εβδομάδα να πάει τον Σεπτέμβριο. Εγώ χαίρομαι που κάναμε το πρώτο βήμα για την απαλλαγή βίζας για τους ε, Κωσοβάρους. Είναι η μόνη χώρα των Δυτικών Βαλκανίων που δεν επιτρέπεται να ταξιδέψουν οι υπήκοοι τους ελεύθερα. Ε, το μήνυμα όμως απευθύνεται και στους πολιτικούς τώρα της χώρας, κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Γιατί δύο πράγματα πρέπει να γίνουν. Γιατί και η Επιτροπή μας και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και η Ολομελία θα υπερψηφίσουν και στο Συμβούλιο θα υπάρχει στήριξη. Και αυτό σημαίνει πως η χάραξη των συνόρων με το Μαυροβούνιο που συμφωνήθηκε πέρσι πρέπει να κυρωθεί από την συνέλευση και ζητώ από τους βουλευτές του Κοσφοπεδίου να το κάνουν και η κυβέρνηση της χώρας πρέπει να προχωρήσει περαιτέρω στις καταδίκες ε, υψηλό βαθμόν για διαφθορά. Γιατί δείξαμε σήμερα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπέρ του να ανοίξει η πόρτα για να ταξιδεύουν οι Κωσοβάροι χωρίς βίζα, αλλά τώρα και αυτοί πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Για να διασφαλιστεί το ταξίδι χωρίς βίζα για τους πολίτες τους. Ε, ευχαριστώ. Σημείο 6. Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι του Ιράν στη συνέχεια της πυρηνικής συμφωνίας. Η κυρία... Α, όχι, ο κύριος Χάουιτ. κυρία Σάκε είναι στην Ίντα υπεύθυνη. Ο κύριος Χάουιτ. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι από τα πιο ενδιαφέροντα με έχουν απασχολήσει στο Κοινοβούλιο. γνωρίζετε ότι οι συνάδελφοι και άλλοι που ασχολούνται με τα δικά μας θέματα ενδιαφέρονται πάρα πολύ και πήγαμε στο Τεχερά, στην Τεχεράνη και είχαμε συνεχθεί πριν τη συμφωνία με την κυρία Μογγελίνη διαδραματίσαμε σημαντικό ρόλο όσον αφορά την οικοδόμηση εμπιστοσύνη και έτσι να μπορέσει να συναυθεί αυτή η πολιτική συμφωνία. Εμεί ω Κοινοβούλιο να διαδραματίσουμε ένα ρόλο. Αυτό προσπαθήσαμε για καλύτερες σχέσεις με την ε, χώρα και να υπάρχει αμοιβαία ωφέλεια στο μέλλον. Συνεργαστήκαμε μαζί με την κυρία Μογκερίνη, όλοι οι συνάδελφοι και τις υπηρεσίες της και το Σαββατοκύριακο θα ξαναπάω στη χώρα για περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων. Και έχουμε σημειώσει πρόοδο ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ε, task force της κυρίας Μογκερίνη και θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο άμεσο μέλλον. Ξέρετε ότι ε, ε, έχω ε, ε, λάβει υπόψη τις επικρίσεις για το Ιράν. πάντως θεωρώ ότι τελικά θα πετύχουμε μια ευρεία συνένεση και ότι τελικά θα έχουμε κάποια διαδικασία ε, επικοδομητική. Αυτό είναι το πνεύμα της έκθεσης. Στο πρώτο τμήμα προσπαθούμε να ορίσουμε το πλαίσιο των σχέσεων που θέλουμε και με ποια διαδικασία θα πετύχουμε αυτές τις σχέσεις. Δεν λέμε ότι ε, από το βράδυ στο πρωί θα έχουν εξομαλυνθεί οι σχέσεις γιατί ε, προηγήθηκε μακρά περίοδος ε, απομόνωσης και τώρα έχουμε και τη σκληρή περίοδο επικοδόμηση εμπιστοσύνη για την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τον αμοιβαίο σεβασμό. Αυτό το προσπάσαν και οι δύο πλευρέ. Θα πρέπει να φυσικά λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν κοινά συμφέροντα. Θα πρέπει επίση να λάβουμε υπόψη τις διαφορές μας, θα πρέπει αυτέ να τις αποτυπώσουμε, να, τις, ε, τους δώσουμε κάποια μορφή και ε, οπότε θα πρέπει να θέσουμε και τα υπέρ και τα κατά της κατάστασης. Επίσης, λέω για το πώς θα βελτιώσουμε τις σχέσεις σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής. Εκεί όπου μπορούμε να τα βρούμε και βέβαια με κάθε σεβασμό στις διαφωνίες μας. Θεωρώ ότι είναι ισορροπημένη εδώ η αποτύπωση των απόψεων όλων των πτερίγων του Κοινοβουλίου, τέλο πάντων μας. Επιτροπή Και λέμε ότι θέλουμε αυτές τις ε, νέε υποδομέ τη εξωτερική υπηρεσία εξωτερικής δράσης τη ΕΕΤ και Κάποια κρατημέλη προσήγησαν τη χώρα και εδώ στο Κοινοβούλιο είπαμε ότι θέλουμε μέσω της έκθεσης να υποστηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες. Επίσης, θέλουμε να υπάρξει κοινοβουλευτική συνεργασία μεταξύ ε, Κοινοβουλίου και της χώρας. Η αντιπροσωπεία μας διατύπωσε στους ε, Ιρανούς συναδέλφους τις προτάσεις μας ότι θέλουμε να υπάρξει κοινοβουλευτικό διάλογο αντιτρομοκρατικού χαρακτήρα. Αυτό είναι κοινό συμφέρον και των δύο πλευρών. Οπότε θα πρέπει να διερευνηθούν οι προσεγγίσεις των δύο πλευρών. Όλα αυτά τα τονίζουμε και θεωρούμε ότι είναι και αυτό ένα βήμα συνεργασίας. Αυτές οι διακοινοβουλευτικές σχέσεις. Τώρα, ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ έχω εργαστεί στην Υποπιτροπή και ήμουν και συντονιστής για την πολιτική μου ομάδα πριν γίνω συντονιστής εδώ. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι είχα αγνοήσει τα προβλήματα. Όμως δεν θέλω να προσπεράσω το θέμα στην έκθεση. και εγώ θέλω κάτι να κάνω να χαϊδέψω τα αυτιά των ε, Ευρωπαίων ακτιβιστών και να ρίξω τους ε, ακτιβιστές που δρούν στη χώρα. Θα πρέπει ομένως κάτι να κάνουμε για να κάνουμε τη διαφορά και να βελτιωθεί η κατάσταση στο Ιράν. Επομένως, ταπεινώς σας προτείνω τις ε, ιδέες μου και παρακαλώ να τις διαβάσετε προσεκτικά γιατί υπάρχουν κάποια ζητήματα που μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο. Ήδη έχει αρχίσει ο διάλογο για τα ανθρωπινά δικαιώματα στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου. Μιλούμε και για την θανατική ποινή, Θεωρούμε να παγώσουν οι εκτελέσει των ανηλίκων. Προσυπέγραψε η Γεράντη σχετική συνθήκη. Επομένως, ε, όλα αυτά συνάδουν με τις διεθνεί υποχρεώσει της χώρα. Και αυτό είναι πρόοδο επίση σε λεπτομέρειε αναφέρομαι στις εκτελέσεις που 80% από αυτές αφορούν καταδίκες σε σχέση με ναρκωτικά. Ε, Οι της αρμόδιες αργίες και ανεγνώρισαν ότι η πολιτική τους δεν αποδίδει. Θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας. Υπάρχει ε, σχετικό νομοσχέδιο που συζητείται όσον αφορά τη μείωση των εκτελέσεων. Οπότε, αν συνεργαστούμε τα θέματα τη ανεργική ποινή και αυτή τη ε, πολιτική των ναρκωτικών, ε, θα ξεκινήσει αυτή η πρωτοβουλία του, του ίδιου του Ιράν. Και έτσι πιστεύουμε ότι θα κάνουμε την διαφορά και θα μειώσουμε τις ε, εκτελέσεις. Αυτό θα είναι πολύ επικοδομητικό και γι' αυτό είπαμε να εστιάσουμε προσοχή μας και αυτό στο θέμα. Εμπόριο και οικονομικά. Έχουμε την σχετική έκθεση της Αρμόδιας Επιτροπής. Έχω συνεργαστεί με την Επιτροπή αυτή και εδώ αναφέρεται ότι είμαστε υπέρ της Ένωσης κάποιες διαδρομές που θα οδηγήσει στον ΠΟΕ τη χώρα. Αυτό ίσως φαίνεται υπερβολικό, αλλά όμως για να φτάσει στον που η χώρα προϋποτίθενται κάποια άλλα διαδήματα, κάποιες άλλες φάσεις που είναι φυσικά σημαντικά. Διαφάνεια, καταπολέμηση της διαφθοράς, επενδύσεις, όλα αυτά που είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης. Γι' αυτό σας λέω ότι και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε οικοδόμηση εμπιστοσύνη μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωσης και Ιράν. Και αυτό επίσης τα θέματα που με σεβασμό θα τα συζητήσουμε επίσης. Έχουμε κάποιους περιορισμούς, κάποιες κυρώσει που έχουν και τραπεζικό χαρακτήρα, οπότε ε, ε, υπάρχει τώρα προσπάθεια να αρθούν αυτοί οι φραγμοί για να υπάρχουν καλύτερε οικονομικέ σχέσει και να ωφεληθούν οι επιχειρήσει των τόσων ευρωπαϊκών χωρών που έχουν εκεί πέρα συμφέροντα. Όμω οι ε, περιορισμοί που έχουν επιβάλει η ΕΠΑ είναι ένας φραγμός. Οπότε γι' αυτό και η κυρία Μογκερίνη συνεργάζεται με τον κύριο Κέρι για να δούμε τι θα γίνει. Τώρα επίσης για τα οικονομικά αναφέρομαι για στις επενδύσεις ποιοτικά και ποιοτικά, κάτι το οποίο παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Τότε που σταμάτησε το εμπάργο είπαμε ότι θα πρέπει τα διεθνή πρότυπα να εφαρμοστούν και στο Ιράν. Επίσης, η συνεργασία σε πολλούς τομείς, να μην σας τα πω τώρα ένα προς ένα, αλλά δεν θέλω τώρα να επαναλάβουμε όσο προβλέπονται στην συμφωνία τα πυρηνικά. Πολλοί θα το θέλανε στην Ουάσινγκτον γι' αυτό και ήταν κατά. Και ε, στην Τεχεράνη κάποιοι είναι κατά αυτή τη συμφωνία. Οπότε και οι Αμερικανοί και οι Πέρσε κατά τη συμφωνία αυτή είναι μειοψηφία. Ίσως και έχουμε και εδώ τέτοιους, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν κάθομαι να αναλύσω την ε, συμφωνία για τα πυρηνικά. Αυτό είναι θέμα της κυρίας Μογκερίνη. Αυτό που κάνω είναι να δούμε τι θα γίνει με, επίσης με τα ανανεώσιμα, νεώσιμες πηγές ενέργειας, ασφάλεια των πυρηνικών, χρησιμοποίηση της πυρηνικής ενέργειας για ελληνικούς σκοπούς, διαχείριση ε, προσφύγων, τεχνολογία, πανεπιστήμια, σχολεία, ε, ανταλλαγές και πολλοί τομείς που είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον του μέσου ανθρώπου. Γι' αυτό θέλουμε την ε, συνεργασία. Και έχουμε εδώ ένα ολόκληρο θεματολόγιο σύμφωνα με τις διαπραγματεύσεις της ΥΠΑ, της εκπροσώπου και του ΙΠΕΞ της χώρας. Και έχουμε άλλωστε και τη σχετική κοινή πρόσφατη ανακοίνωση. Στο τέλος λέμε για τον περιφερειακό ρόλο της χώρας. Και συμφωνώ με τον κύριο Μπροκ. Δεν αποκρύπτουμε και έχουμε βασικό κίνητρο για αυτή την έκθεση το ότι εάν μπορούμε να συνεννοηθούμε υποδομητικά με τη χώρα αυτό θα είναι αποφασιστικό στο να φρενάρουμε τα όσα γίνεται σε Ιεμένη, Λιβύη, Συρία και γενικότερα την αστάθεια στην περιοχή όπως ας πούμε την αστάθεια του Λίβανου. Μπορεί να πείτε ότι όλα τα λέμε εδώ στρογγυλά. Δεν είναι έτσι. Ο καθένα. έχει τι ιδέες του, και φυσικά δεν μπορούν να σταματήσουν πολύ, αλλά λέω ότι αν κάτι στο τραπέζι να πραγματεύσουν το Ιράν και αν συνοηθούν με τη χώρα, ε, τότε υπάρχει μια ευκαιρία να σημειωθεί κάποια πρόοδο σε αυτού όλου του περιφερειακού πολέμου και συγκρούσει. Είμαστε περήφανοι για αυτό που κάναμε. Και όσον αφορά την ε, θέση μου για το Παλαιστινιακό, ναι, θέλω μια λύση δύο χωρών στο Παλαιστινιακό. Θέλουμε ασφάλεια και ειρήνη για όλους και όπως λέω για όλους χωρίς εξαίρεση το γράφω στην έκθεση έχει πολλούς ε, Εβραίους στο Ιράν και αυτοί έχουν συμφέρον επομένω, για αυτή την υπόθεση της ειρήνευσης στην περιοχή πολύ προσεκτικά έχω κάνει τις διατυπώσεις μου και να το λάβουν αυτό η υπόψη όσοι είναι φιλίποπτη προς το Ισραήλ. Θα έχουμε και τροπολογίες, φυσικά έπρεπε η έκθεση να έχει συγκεκριμένο μήκος και θα ακούσω μεγάλη προσοχή τις απόψεις για όλα τα επίμεγα σημεία της έκθεσης. Και θα προσπαθήσω να συνεργαστώ με όλες τις πολιτικές ομάδες και να βγάλουμε όσο γίνεται καλύτερη έκθεση. Και επομένω με αυτό το πνεύμα θα κάνω την επίσκεψή μου στη χώρα το Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ το Ιράν ενδεχομένω ε, να γίνει ένα σημαντικό σύμμαχος. Ο κύριος Πρέντα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο Χάουιτ για την παρουσίαση και για το ενδιαφέρον που έχει δείξει στο θέμα αυτό. Το θέμα της στρατηγικής μας ε, μετά την ε, συμφωνία είναι πάρα πολύ σημαντικό ασφαλώς και κατανοώ τους οικονομικούς και εμπορικούς ε, λόγους τις οποίες μας παρουσίασε ο Ρίτσαρτ και τους ε, γεωπολιτικούς λόγους που θα πρέπει να λεφτούν υπόψη για να υπάρξει μεγαλύτερη δέσμευση με τη χώρα αυτή. Και προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να επιδείξουμε μεγαλύτερη σοφροσύνη. Ακούσαμε τον συνάδελφο, ο οποίο ήταν σχεδόν παθιασμένο όταν μα μίλησε. Όταν συζητήσαμε πριν από ένα χρόνο στην ε, Ολομέρεια τα θέματα των πυρηνικών, είχαμε εκφράσει ήδη ε, την ελπίδα να υπάρξει ε, μια αλλαγή σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, να υπάρξει μια μεταρρύθμιση και εκεί. Αυτό πριν από ένα χρόνο. Έχει περάσει λοιπόν πλέον ένας χρόνος και πρέπει να διαπιστώσουμε ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Οι εκτελέσεις το 2015 στο Ιράν ήταν ε, πιο πολλές από ποτέ. Και η κατάσταση των γυναικών έχει επιδεινωθεί, η Βασανιστήρια μαστιγώσεις ε, επίσης στην καθημερινή διάταξη. Και ο Ρίτσαρντ είναι, ήταν υπεύθυνο για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο με απασχολεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Αθηναντική ποινή, δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό που ορίζει η παράγραφος υπαριθμών 5, καθώς ε, δεν πρόκειται για απόκληση απόψεων η αντίθεσή μα ε, στη θανατική ποινή αποτυπώνει τι βασικές αξίε τις οποίε ε, αντιπροσωπεύουμε. Αυτό θα πρέπει να επικαλυστούμε. Δεν πρόκειται για μια απλή διάσταση απόψεων προ Θεού. Στην παράγραφο 7 τώρα αναφέρεται ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούμε ε, συμφωνίες πλαίσιων. Στο 18 μιλάμε για την απελευθέρωση από τις θεωρήσεις για μια κατηγορία ατόμων, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν παράλληλα όμως και εγγύησεις για ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι ανταπισμένος, δε, ότι δεν θα πρέπει να κλείνουμε τα μάτια σε όλα αυτά λόγω της πυρηνική συμφωνίας. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να απαιτούμε βελτιώσεις ε, σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και άρα θα ήθελα λοιπόν να υπάρξει μια αναπροσαρμογή της συμφωνίας για να τονιστεί το θέμα των δικαιωμάτων. Αυτό λοιπόν με απασχολεί και έχω καταθέσει πάρα πολλές τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή και άλλωστε Έχουμε ζητήσει επανειλημμένοι από τους σοσιαλιστές φίλους μας να μιλάνε και για το Ιράν, όχι μόνο για την Σαουδική Αραβία, γιατί είναι πολύ επικριτική σε ό,τι αφορά την Σαουδική Αραβία, αλλά επιδεικνύουν έτσι πιο φιλική διάσταση ε, σε ό,τι αφορά τους Ιρανούς. Και θεωρώ ότι αυτό είναι προβληματικό σε ό,τι αφορά και τους Ιήτες του Ιράν. I think we have to be a little... Ο Πρόεδρος, ε, να είμαστε και λίγο πιο σύντομοι, γιατί στις 9 θα έρθει και η κυρία Μογκερίνη. Και έχουμε ακόμα 10 άτομα στο κατάλογο των ομιλητών. Ο κύριος Λίτς. Ε, κοιτάξτε, δεν θα γρηγορέσω. Να τονίσω την κατάσταση, να ευχαριστήσω και τον Ριτσάρτ και τον κύριο Πρέντα που έτυξαν το θέμα της εθαντικής ποινής. Χίλια άτομα. Χίλια άτομα βρέθηκαν σε αυτήν την κατάσταση πέρσι στο Ιράν. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό. Ακόμα και οι Ιρανοί στη Γερμανία το έδειξαν το θέμα αυτό. Ακόμα και οι δημοσιογράφοι. Σίγουρα λοιπόν θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ, κύριε Τάνοκ. Η κυρία Φωτίγκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις να κάνω, επιτρέψτε μου. εκτελέσεις, καταρχάς. Όχι μόνο τα αριθμητικά στοιχεία, αλλά και η δυναμική του όλου θέματος. Σε ό,τι αφορά αυτό, το, αυτό που καλούμε να μετριοπαθές καθεστώς στο Ιράν. Σημειώθηκε αύξηση όμως. Και αυτό είναι προβληματικό. Σημαντικό πρόβλημα για μένα. Δεύτερο, το θέμα της περιφερειακής ασφάλειας. Και εδώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ποιος είναι ο ρόλος του Ιράν, θεωρείτε, στην υποστήριξη του Ασάντ. Ποια είναι η επιρροή στο συριακό ζήτημα και πώς θα μπορούσε να επιληθεί η συριακή κρίση με τη συμβολή και κατά δεύτερον ο ρόλος τους στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η στάση που τηρούν έναντι οργανώσεων όπως η Χαμάς και ενδεχομένω η προθυμία του Ιράν να συμμαχίσει μαζί μας στην καταπολέμηση αυτών των οργανώσεων. Ευχαριστώ κυρία Σχάκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον Ρίτσαρτ για τη δουλειά που έχει κάνει για το θέμα αυτό και δυστυχώς ε, μένα καλούμαστε να αντιδράσουμε στην Ειρηνική Συμφωνία, αλλά δεν θα κάνουμε, καλή αργά παρά ποτέ. Εγώ στην ΙΝΤΑ έχω επικεντρωθεί στα θέματα τα εμπορικά. Δεν θα τα αναφέρω τώρα, αλλά ως Κοινοβούλιο θεωρώ ότι είναι σημαντικό να παίξουμε το ρόλο μας για να υπάρχει μια ευρεία ατζέντα με το Ιράν, αλλά να μην είμαστε και αφελείς. Το σύστημα στην Ισλαμική Δημοκρατία περιλαμβάνει ε, μία αντίθεση μεταξύ των συντηρητικών και των ακτιβιστών και αυτό οδηγεί σε προβλήματα έλλειψη ε, δημοκρατίας, ε, ελευθερία έκφρασης, κάτω δικαίου, ύστερα έλλειψη δυτικοποιήσεων. Συνεχίζεται να υποστηρίζεται το Ασάντο, ο οποίος βομβαρδίζει του ίδιου τον του λαού. Και έχουμε κάνει τρεις ε, αποστολές ε, από πλευρά της Επιτροπής μας και έχει καταστεί σαφές το πόσο βαθιές είναι οι ρίζες του προβλήματος και από την άλλη και πόσο απόλυτα απαραίτητο είναι να επικεντρωθούν στο ανθρώπινο κεφάλαιο που είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο της χώρας ε υψηλή εξειδίκευση και κατάρτιση και εκπαίδευση. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να επανασυνδεθούν με τον κόσμο, αλλά απομονώνται Μιλήσαμε για τι εκτελέσει, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να τονίσουμε και τα δικαιώματα των γυναικών, τη ελευθερία έκφραση, του τύπου κτλ. Υπάρχουν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. Αυτό δίνει μια ευκαιρία συνεργασία, καθώ και οι ενεργειακέ πολιτικέ. Άρα, εγώ διακρίνω και σοβαρές, ε, σοβαρά προβλήματα θα πρέπει να επιληθούν, αλλά και πολλές ευκαιρίες. Να μην είμαστε αφελείς και να είμαστε ρεαλιστές. Αυτό συστήνω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συμφωνία του περασμένου Ιουλίου και η άρση των κυρώσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα έβγαλαν το Ιράν από την απομόνωση που του είχε επιβάλει η Δύση. Περιμένουμε λοιπόν από το Ιράν να αξιοποιήσει επικοδομητικά τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει όχι μόνο στη Μέση Ανατολή αλλά και στην παγκόσμια οικονομία, συνεισφέροντας την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη. Από αυτή την άποψη, η συμμετοχή του Ιράν στην επίλυση των διαφορών συγκρούσεων και πολιτικών κρίσεων είναι σημαντική και νομίζω ότι θα πρέπει να κρίνεται συνεχώς. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή οξύνεται καθημερινά και οι συγκρούσει προσλαμβάνουν φιλετικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά, με ορισμένου παράγοντε στην περιοχή να κάνουν χρήση των θρησκευτικών διαφορών για την υποκίνηση πολιτικών κρίσεων και πολέμων μυσαλλοδοξία με σκοπό, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση του ελέγχου στην περιοχή. Σήμερα, έπειτα από μια μακριά δύσκολη περίοδο για τι σχέσει του Ιρανικού λαού με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναπτύσσεται ένα φιλόδοξο, πολυεπίπεδο, διατομιακό διάλογο σε κλίμα οικοδόμηση αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμού στη βάση τη αξιολόγηση των κοινών συμφερόντων και διαφορών κατά τρόπο που να ωφελεί τόσο τον ιρανικό λαό όσο και τον ευρωπαϊκό. Σε αυτό το διάλογο νομίζω ότι έχουμε χρέο σαν ευρωβουλευτέ να δουλέψουμε ώστε να αναπτύξουμε την κοινοβουλευτική διάσταση μεταξύ των σχέσεών μα με το Ιράν. Θα ήθελα ειλικρινά να συγχαρώ τον κύριο Χάουιτ για τη δουλειά που έχει κάνει, παρουσιάζοντα μια ισορροπημένη έκθεση που απαντά στι περισσότερε από τι προκλήσει τη παραπέρα ανάπτυξη των σχέσεών μα με το Ιράν. Ωστόσο, κλείνοντα, θέλω να επισημάνω την έλλειψη ισχυρών αναφορών σε εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά τις γυναίκες, τις μειονότητες κλπ το Κοινοβούλιο ακριβώ πάνω σε αυτή την επικοδομητική βάση διαρκού συνεργασία και διαλόγου που αναφέραμε, θα πρέπει να εκφράσει για μια ακόμη φορά την ειλικρινή του άποψη, χωρί καμιά διάθεση για εσωτερικέ παρεμβάσει, αλλά να διασφαλίζει τη σχέση αυτή και να βασίζεται στον εμβαίο σεβασμό των διεθνών προτύπων και αρχών. Εκ μέρου λοιπόν τη ΓΚΟΕ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να θα καταθέσω τροπολογίε για τη βελτίωση τη έκθεση και θα στηρίξω πολλά σημεία που πιστεύω ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Χάουιτ για την πρότασή του. Περιέχει, όπως είπαμε, πολλές σημαντικές πτυχές, αλλά βεβαίως θα καταθέσω τροπολογίες ε, για την ομάδα μου. Ε, μας μας ενδιαφέρει κυρίως ενισχυμένη συνεργασία με το Ιράν στην προστασία, παραδείγματος χάρη, του περιβάλλοντος και στην περιβαλλοντική τεχνολογία. Εδώ νομίζω μπορούμε να πτύχουμε πολλά προς αμοιβαίο όφελος και να βοηθήσουμε ιδιαίτερα με τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ιράν, ειδικά σε κάποιες ε, λίμνες. Σημασία έχει επίσης η ενεργειακή πολιτική που πρέπει να αναδιαταχθεί τελείως στο Ιράν. και βεβαίως πρέπει να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω λοιπόν πως ε, στο Ιράν ή στις σχέσεις ε, μεταξύ μας έχει υπάρξει μια σοβαρή αλλαγή. Τις ε, πρώτες φορές είχαμε μια γενική άρνηση όταν θίγαμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εν τω μεταξύ έχει αλλάξει η στάση και τα συζητάνε. Νομίζω πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την αλλαγή. Νομίζω πως μπορούμε εδώ πέρα να επιτύχουμε αρκετά πράγματα αν ε, αναφερθούμε σε συγκεκριμένα ζητήματα. Αναμένω λοιπόν τη συνεργασία με τους ε, συναδέλφους και είμαι σίγουρος πως θα καταλήξουμε σε μια λογική έκθεση. Ευχαριστώ. Ε, ε, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω πολωνικά. Κοιτάξτε, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ισορροπία στον ε, μουσουλμανικό κόσμο. Οι ΣΥΙΤΕΣ είναι μειονότητα και εάν υποκύψει το Ιράν σε αυτά τα οποία θέλουμε, ίσως ε, στραφούν εναντίον του οι υπόλοιποι μουσουλμάνοι και οι Σουνίτες ε, και έτσι μπορεί να επιδεινωθεί η κατάσταση στη Συρία. Ίσως πέσει ο Ασάντ και τότε χιλιάδες χριστιανοί και αλεβίτες θα πρέπει να φύγουν και να έρθουν στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να σεβόμαστε τις μειονότητες μεταξύ των οποίων και οι Συΐτες που είναι μειονότητα στον Ισλαμικό κόσμο. Ευχαριστούμε. Richard Χάουιτ είναι αξιόλογη η έκθεση και είναι μια προσέγγιση που είναι σωστή, την έκανε για άλλη μια φορά, αυτή τη βαθμία δηλαδή προσέγγιση με τη χώρα και είναι σαν το ε, ε, εκρεμές ε, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή από εκεί που ήταν κράτος παρείας τώρα θα είναι εταίρος. Δεν είναι όμως παρείας, είναι πολύ σημαντική η χώρα για την περιφέρεια αλλά βέβαια ακόμα δεν είναι φυσιολογικό εταίρο. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει μια έξομάλυση των σχέσεων κατά ε, φάσει, θα πρέπει να προσέξουμε όπω είπατε και πρώτα πρώτα βέβαια προϋπόθεση είναι να υλοποιήσουν 100% ε, όπως θα μας πει και η κυρία Μαγκερίνη τη συμφωνία για τα πυρηνικά. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ισχύσει αυτή η προϋπόθεση. Και τώρα πιο πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να προσέξουμε τη στρατιωτικοποίηση της περιοχής ακριβώς όπως αναφέρατε στην παραγραφό 20 αν δεν κάνω λάθος ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη βέβαια το ότι είναι τώρα πιο ευέλικτη για τα πυρηνικά για αυτή η καινούργια προσέγγιση της χώρας από την άλλη μεριά να μην οδηγήσει σε σκληρή προσέγγιση όσον αφορά τα, τα βαλιστικά όπλα τα οποία αναπτύσσει η χώρα και αυτά, αυτό είναι λόγος να ανησυχεί κανείς για το τι γίνεται στην περιοχή τώρα. Να προσέξουμε και για την Συρία, γιατί εγώ θέλω οπωσδήποτε να κάτσει στο τραπέζι το Ιράν. Είναι παράλογο να συζητούμε χωρίς το Ιράν το Συριακό. Οπότε ακριβώς γι' αυτό η μέχρι σήμερα εμπλοκή της χώρας για αυτές τους, τις διεθνείς ε, πλατφόρμες, τα διεθνή φόρα, δεν έχει αποδώσει ιδίως όσον αφορά ε, ε, Task Force, όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, δεν έχουν συμβάλει οι Ιρανοί μέχρι τώρα Άρα να είμαστε ανοιχτοί, αλλά να είμαστε και προσεκτικοί. Uh, thank you, Chair. Uh, can I also welcome uh, Καν. Μπράβο στον Ρίτσαρτ για όσα έκανε για την ε, έκθεσή μας. Είναι πολύ σημαντική γιατί είναι και η χώρα σημαντική και άρα ας εξασφαλίσουμε υγιές με ενδιαφέρουν όλα αυτά που είπε ο Ότι δηλαδή όλη η περιοχή να θεωρήσει ότι τα πράγματα έχουν πάρει τη σωστή ρόντα στις σχέσεις μας. Βεβαίω και μπορεί να παίξει θετικό ρόλο το Ιράν στο Συριακό. Άρα και εμείς να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας αναλόγως με το Ιράν. Και να δούμε και τι θα γίνει και με την δυσκευτική βία, που είναι ακόμα ένας προβληματικός τομέας στην περιοχή. Έχουμε κλιμάκωση αυτής της κρίσης. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτό το πρόβλημα για τελευταίες εβδομάδες. Είδαμε πόσες ζωές έχουν χαθεί. Και για τα ανθρώπινα δικαιώματα επίσης δεν μπορώ από τίποτα κατά των θέσεων του Ρίτσαρντ. Ξέρω τι έργο έχει επιτελέσει το παρελθόν και συμφωνώ με την προσέγγιση του, αλλά α εξασφαλίσουμε η προσέγγιση μας να έχει κάποια συνέπεια και να μην καταλήξουμε σε δύο μέτρα και δύο σταθμά σε σχέση με τα άλλα μέτωπα που έχουμε ανοίξει σαν Ένωση. Συνεργασία σε πολλούς τομείς. Ναι, έτσι τελικά θα ενδυναμωθεί η σχέση μας με τη χώρα. Οπότε θα υπόλοιπε και και θα προχωρήσουμε την υπόθεση. Thank you, Chair. Uh, two quick points, first of all. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο γρήγορα σημεία. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το πολύ καλό κείμενο με το Ιράν. Και τον κύριο Πρέντα ευχαριστώ γιατί υποστήριξε ένθερμα τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή. Συμφωνούμε, συμφωνούμε. και θα περίμενα να ε, έχει την ίδια στάση και για άλλε γειτονικέ χώρε, από την Παρτιατική Ασία, όταν κάνουμε ε, σύμφωνε εταιρική για παράδειγμα. Επίση, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει πλέον και μία μόνιμη αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ιράν, γιατί πώ θα προτείνουμε επίση ε, συμφωνία σχέσει σχέση αν δεν έχουμε μόνιμη αντιπροσωπεία. Αυτό θα βοηθούσε σίγουρα. Ευχαριστώ. Τεχνική παρατηρήση, Πρόεδρε. Όταν έχουμε περιορισμένο χρόνο, τι δίνουμε στον εισήγητη τόσο πολύ χρόνο και περιορίζουμε τόσο πολύ τον χρόνο για τους υπόλοιπους ομιλητές. Τέλος πάντων, ευχαριστώ. Δεν είναι ισορροπημένη η έκθεση. Ε, δεν τηρεί και τη γραμμή μας για την εξωτερική πολιτική. Δεν θα πρέπει να αγνοούμε και να είμαστε επίοικείς με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις, το θέμα των δημοκρατίας. Ε, γιατί τίφεται στο επίκεντρο η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διατηρήσουμε το πνεύμα των διαπραγματεύσεων για να ωφεληθεί ο κόσμος και στο Ιράν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά στην ε, διπλωματία χρειάζεται αμοιβαιότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση καλά θα κάνει να θυμάται ότι παραμένει το Ιράν ένα θεοκρατικό καθεστώς το οποίο υποστηρίζει τη πολλά και το Συριακό καθεστώς και άλλες τέτοιες ενοπλές ομάδες. Κατά δεύτερον, ζητείται η ανάπτυξη των κοινοβουλευτικών σχέσεων με το Ιράν. Αγνοούνται βέβαια κατάφορα ή πολλαπλέ ε, περιπτώσει παραβιάσεων ανθρώπινων δικαιωμάτων στι πρόσφατε εκλογέ. 60% ε, των ε, καταχωρισμένων εκλογέων α, δεν μπόρεσε να ψηφίσει. Δεν είναι δημοκρατικό το κοινοβούλιο του Ιράν, άρα κατά τρίτον. Η έκθεση δεν αναγνωρίζει καν σχεδόν τι διαφορέ που υπάρχουν μεταξύ Ιράν και Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρήση τη θανατικής καταδίκη. Αυτό είναι, τι να σα πω, τουλάχιστον ε, υπερβολικό στην διατύπωσή του. Τα τελευταία τρία χρόνια οι εκτελέσει έχουν ξεπεράσει τι εκτελέσει των 25 χρόνων πριν και συνεχίζει στου ίδιου ρυθμού και εκτελεί και ανηλίκου στο Ιράν. Κατά τέταρτον, αναφέρεται στην έκθεση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σκοπεύει να αναμειχθεί στα εσωτερικά, αλλά βασίζεται στην αμοιβαία αναγνώριση βάσει των διεθνών προτύπων. Φυσικά, σε αυτά τα πρότυπα συγκαταλέγονται και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Μάρτιο του 2015, ο Αχμήν Σαχμέλ, ο οποίο είναι υπεύθυνο των ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, ανέφερε ότι επιδεινώθηκε η συνολική κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν. Πέμπτον, η έκθεση αναφέρει ότι υποστηρίζεται η επιθυμία του Ιράν να συμμετάσχει στον ΠΟΕ. Αναφέρεται όμω πουθενά είναι έκθεση ότι οι Αλκούτς, οι στρατιωτικοί ε, έχουν στα χέρια τους την βιομηχανία του Ιράν. Γενικά η έκθεση ζητάει καλή θέληση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το καθεστώς είναι αυτό που είναι υπεύθυνο για όσο τραβάει ο λαός στο Ιράν. Ζητάει την καταστροφή του Ιράν, καταπιάζει τον ίδιο τον λαό του Ιράν τα τελευταία 35 χρόνια. Μήπως τα πράγματα θα έπρεπε να είναι αντίστροφα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας ε, κάνει τις περισσότερες ε, εκτελέσεις. Βεβαίως, κατά κεφαλήν και αναλογικά είναι το Ιράν. Πέρσι ήταν σχεδόν χιλιά άτομα. Οι δημόσιες εκτελέσεις κρεμάνε κόσμο από γερανούς τώρα τελευταία είναι η αγαπημένη τους μέθοδος και ειδικά με τους γερανούς φαίνονται και από μακριά οι άνθρωποι. Και εγώ θα ξεκαθαρίσω στον συγητή ότι η έκθεση δεν είναι ισορροπημένη και θα υποβάλω και τροπολογίες για να γίνει πιο ισορροπημένη. Αναγνωρίζω ότι μπορεί να είναι σταθεροποιητικός παράγων στην περιοχή το Ιράν. έχουμε νομίζω μέχρι την μία η ώρα στις 14 του μηνός για να αποβάλουμε τροπολογίες, οπότε υπάρχει ακόμα χρόνος για τους υπερασπιστές ανθρωπινών δικαιωμάτων. Ναι, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Ρίτσαρτ Χάουιτ για το... Εδώ είμαι. Για το σχέδιο έκθεσης. Είναι αφενός σωστό να δούμε ολόκληρο το δυναμικό της συνεργασίας και εκεί πέρα πραγματικά παρουσιάσατε όλες τις πτυχές. Υποστηρίζω οπωσδήποτε το θέμα του ανοίγματο μιας αντιπροσωπείας της Ένωσης, αλλά θα επαναλάβω και αυτό το που είπαν και άλλοι συνάδελφοι για το να είναι ισορροπημένη η έκθεση συνολικά. Πριν από 15 χρόνια είχα συντάξει μια τέτοια έκθεση και είχαμε μια παρόμοια κατάσταση. Είχαμε έναν μεταρρυθμιστή πρόεδρο, τον Χαταμή, και μια εθνοσυνέλευση ανάλογη, με ανάλογη σύνθεση και υπήρχε μια προσεκτική, μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Βεβαίως ξέρουμε ότι άλλαξαν τα πράγματα 2004 δεν επετράπει στους μεταρρυθμιστές υποψηφίους να κατέβουν στις εκλογές και είχαν ανταυτού κατέβει σε απεργία πείνας. Και πρέπει ακριβώς να δούμε αυτή την διαφορά μεταξύ επισήμων και ατύπων δομών στην χώρα. Υπάρχει δηλαδή σύνταγμα πρόεδρος, εθνοσυνέλευση, αλλά υπάρχουν και αυτοί που έχουν την πραγματική εξουσία. Και πρέπει να τους αναφέρουμε. Επίσης ε, και τα 120 θρησκευτικά ιδρύματα τα οποία ελέγχουν την οικονομία. Αυτοί λαμβάνουν τις αποφάσεις. Δεν είναι ακριβώς και συμβατά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Α, πρέπει να τα πούμε λοιπόν αυτά. Thank you. Very much. Ε, σας ευχαριστώ. Συμφωνώ πολύ με την προσέγγιση των συναδέλφων Πρέντα και Σάκη και των άλλων. Εκτιμώ την προσέγγιση του Ρίτσαρντα με την καλή θέληση και τις ελπίδες, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω πως πρέπει να είμαστε ψυχρεμοί και να μην βιαζόμαστε, να μην προτρέχουμε. Νομίζω πως ο ε, συνάδελφος Νταζάν ότι αυτό το οποίο είπε ότι το Ιράν δεν είναι κανονικός εταίρος πρέπει να μας καθοδηγεί γιατί το καθεστώς δεν έχει αλλάξει. Αυτό είναι γεγονός. Ε, και υπόθηκε άλλωστε. Μόλις το προηγούμενο βήμα το Υπουργείο Εξωτερικών τον ΙΠΑ στην έκθεση του για την Παγκόσμια Τρομοκρατία περιέλαβε το Ιράν ε, στις χώρες που χρηματοδοτούν την τρομοκρατία. Και νομίζω πως η βασική προσέγγιση πρέπει να είναι ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και βεβαίως η πλήρωση των όρων της πυρηνικής συμφωνίας πρέπει να είναι προϋποθέσεις για συνεργασία με το Ιράν. Έτσι πρέπει να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη. Μέχρι τώρα το Ιράν ε, και οι κινήσεις του δεν είναι αξιόπιστες. Ε, για τη θανατική ποινή τώρα που αναφέρθηκε. Η παράγραφος 5 αναφέρθηκε. Σήμερα καταδικάζουμε τον Μπαχρέιν. Επειδή εισάγει τη θανατική ποινή. Δηλαδή, αν είναι να μιλάμε για δύο μέτρα και δύο σταθμά, εδώ τα βλέπουμε στην παράγραφο 5 που αναγνωρίζουμε τις διαφορές στην προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιράν. Δηλαδή τους δικαιολογούμε ότι τους εκτελούν, εκτελούν ξέρω εγώ τους εμπόρους ναρκωτικών γιατί τίποτα άλλο δεν μπορεί να γίνει. Κλασική προπαγάνδα ολοκληρωτικού καθεστώτος και οι οικονομικές σχέσεις πρέπει να αποκατασταθούν ε, όταν το Ιράν συμμορφωθεί με τις συστάσεις της ε, ομάδας δράσης του ΟΣΑ, της Financial Action Task Force και βγει από τη μαύρη λίστα. Αυτά και αναμένω και τη συνεργασία με τον εισηγητή. Σας ευχαριστώ. Να κάνω και εγώ κάποιες παρατηρήσεις ως εκπρόσωπος ε, του ΕΛΚΑ, όπου και παίζει το ρόλο και του Σκιώδους εισηγητή, καταρχάς, θεωρώ ότι από πλευράς της ευρωπαϊκής ε, πλευράς θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ε, είναι αξιόπιστη η στάση σε ό,τι αφορά τη σύναψη της συμφωνίας. Και από τη δική μας πλευρά και από τη δική τους πλευρά. Να μην δεθούν λάθος εντυπώσει. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχιστούν τα μέτρα για την οικοδόμηση μια σχέση εμπιστοσύνη και θα πρέπει να κάνουμε και τους απαραίτητους ελέγχου. Βέβαια, δίκιο είχε και αυτός που είπε ότι για την ε, επίλυση της κρίσης ε, της Συρία, στο Ιράκ και για να ε, σταματήσει αυτός ο πόλεμος δια αντιπροσώπου, χρειάζεται και βοήθεια του Ιράν. Θα πρέπει να συμμετάσχει και το Ιράν όλοι αυτοί οι πόλεμοι για το, στη Μέση Ανατολή και με τα προσφυγικά κύματα τα οποία συνεπάγονται. Όλα αυτά θα μπορούσαν να επιληθούν μόνο εφόσον θα διαδραματίσει επικοτινικό ρόλο και το Ιράν. Αυτό ισχύει και για τη Σουδική Αραβία και για άλλους που βρίσκονται από την άλλη πλευρά. Και αν δεν ε, επιλύσουμε την κατάσταση θα έχει αυτό συνέπειες σοβαρές για μας. Τώρα, κοιτώντα την συζήτηση που διεξαγάγεται στο Ιράν και τη στάση του Ιράν, διαπιστώνω ότι δεν είναι θετικό αν τους κυνηγάμε και πάρα πολύ γρήγορα. Δεν θα το εκτιμήσουν. Θα πρέπει να έχουμε ένα ανοιχτό πνεύμα, αλλά και να διατηρήσουμε μια αλφα αξιοπρέπεια. Ιδάλλως αυτό μπορεί να προκαλούσε, ξέρετε, παρανοήσεις. Ο Υπουργός Οικονομικών ε, της Γερμανίας και όχι μόνο αυτός, τρεις ημέρες μετά την υπογραφή της ε, συμφωνίας έκανε τις δηλώσεις έκανε τις δηλώσεις που έκανε, θεωρώ ότι δεν ήταν θετικό αυτό, ούτε μας βοηθάει στη στάση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης να το πω και εγώ, όπως το είπαν και άλλοι, ότι πρόκειται για μια διχασμένη ε, χώρα σε ό,τι αφορά το πολιτικό σύστημα, το θρησκευτικό τμήμα. Εξακολουθεί να υπάρχει ο πρόεδρος Ρουάν και η εκλογή του, καθώς και τα, οι άλλοι ηθήνοντες θεωρώ ότι από πλευρά κρατική ε, πετύχαμε μία αλφα, έναν αλφα ανοιχτό χαρακτήρα. Και αυτό γιατί η χώρα χρειάζεται συνεργασία αν θέλει να διατηρήσει το επίπεδο που έχει στο κόσμο, στο, στο λαό του, με υψηλή εκπαίδευση μεταξύ των νέων κτλ. Και να παρατηρήσουμε ότι για μας αυτό αποτέλεσε μια ευκαιρία το γεγονός ότι δεν ε, προετοιμάζουν πυρηνική βόμβα. Και φυσικά αυτό οδηγεί σε μια συζήτηση ότι αν δεν τηρηθούν οι προδιαγραφέ για τα πυρηνικά θα επανέλθουν οι κυρώσει. Και θεωρώ ότι αν δεν υπήρχε αυτός δυνατότητα θα άλλαζε η κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό το εργαλείο, αλλά να επιδιώξουμε λύσεις βάθμιες και σταδιακές, όπως έχει γίνει φέτος. για να δημορφωθεί με πιο θετικό και επικοδομητικό τρόπο όλη η περιοχή. Να προσέξουμε τώρα με το Κοινοβούλιο τίθεται το θέμα ενός ε, λαού που έχει σε μεγάλο βαθμό θεοκρατικές στάσεις; Η εκλογή κάποιων ευθύνοντων ήταν αρκετά ελπιδοφόρα. Δεν μπορεί να βγει υποψήφιο οποιοδήποτε. Γιατί το θεοκρατικό κομμάτι δεν δέχεται πολλούς και πολλούς προοδευτικούς δεν τους δέχεται καν. Και αυτό αποτελεί φυσικά και την άλλη όψη του νομίσματος. Έχουμε πλεονεκτήματα, έχουμε και μειονεκτήματα. Και Ρίτσαρτ, και εγώ θα ήθελα να αναπτύξουμε ε, σχέσεις με το Κοινοβούλιο. Δεν θα ήθελα όμως να μεταβούμε εκεί ως Κοινοβούλιο. Γιατί έχουμε επισκεφτεί την περιοχή. Είναι η σειρά των Ιρανών να μας επισκεφτούν. Θα μπορούσαμε λοιπόν να απευθύνουμε μια νέα πρόσκληση στο νέο κοινοβούλιο για να μας επισκεφθούν ε, στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο. Γιατί θεωρώ ότι δεν θα σωστό να πάμε εμείς δύο φορές συνεχόμενες. Θα πρέπει να υπάρχει μια αλφα σειρά και μια αλφα ισορροπία. Σας ευχαριστώ πολύ και το λέγω να πάρει ο συγγετής. Α, συγγνώμη, ο κύριος έχει ζητήσει το λόγο επίσης. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. η συζήτησή μας έχει ε, επικεντρωθεί ε, υπερβολικά και χωρίς λόγο τόσο πολύ στην θρατική καταδίκη. Γιατί αυτό στο οποίο θα πρέπει να επικεντρωθεί η έκθεση αυτή είναι οι θεμητές ε, ανησυχίες περί ασφάλειας του Ισραήλ. Είναι βασικό να μην αποτελεί πηγή αντισημιτικής προπαγάνδας στο Ιράν. Και επίσης θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι οποιαδήποτε έκθεση αναφορικά με την ασφάλεια στην γενικότερη περιοχή θα πρέπει να διατυπώνει ρητά ότι το Ιράν θα πρέπει να δρά βάσει καλής πίστης. Αυτά τα πράγματα δεν θα πρέπει να τα υποδεικνύουμε ή να υπονοούνται. Θα πρέπει ρητά να αναφέρουμε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να σωπαίνουμε για τέτοια ζητήματα. για τόσο πολλά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και η επεκτατική τάση του ΝΤΑΕΣ, το Ιράν θα μπορούσε να αποτελέσει αντίβαρο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν προβλήματα και οι φίλοι μας θα μπορούσαν να βρεθούν σε κατάσταση κινδύνου. Θα πρέπει λοιπόν προ καταρχικά θα πρέπει εκ των προτέρων να αντιμετωπίσουμε και να σκεφτούμε τα προβλήματα αυτά και να πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Γιατί είναι θανατική καταδίκη, θα πρέπει να γίνει σεβαστό το δίκαιο, αλλά να έχουμε υπόψη ότι στι ΗΠΑ επίση υπάρχει θανατική καταδίκη. Και δεν ασκούμε κριτική στι ΗΠΑ για τη θανατική ποινή. Όχι με τον ίδιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Να επικεντρωθούμε λοιπόν στα ζητήματα τα οποία απειλούν την ανθρώπινη ζωή. Ο ρόλος και η στάση του Ιράν έναντι του Ισραήλ και τη Χεσμολά. Να μην επικεντρωνόμαστε περιβολικά σε δευτερεύοντα ζητήματα. Και κάτι άλλο. Είναι λυπηρό το ότι ο ρόλος του Ιράν στο, στον πόλεμο της Συρίας έχει αυξηθεί. Αλλά και εμείς έχουμε ε, συμβάλλει σε αυτόν τον πόλεμο. Ο κύριος έχει κάνει το δικό του κομμάτι. Ευχαριστώ. Κύριος Χάουιτ. Ευχαριστώ. Έκανα μια ξεκάθαρη δήλωση. Τώρα μια που έρχεται και η πατία εκπρόσωπος θα είμαι σύντομος για τον κύριο Πρέντα. Ναι, γνωρίζω ε, πιθανό πρόβλημα και διάλεξα πολύ προσεκτικά τις λέξεις μου και μάλιστα μιλάω για τα θεμητά συμφέροντα ασφαλείας των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και του Ιράν ε, και των άλλων χωρών και ότι η περιφερειακή δομή ασφαλείας θα είναι ένας να καταπολεμηθούν οι συγκρούσεις. Και συμφωνώ με τα σχόλια του συναδέλφου του κυρίου Χάν ότι πρέπει να δοκιμάσουμε την αποκλιμάκωση μεταξύ Ριάντ και Τεχεράνης και αντιλαμβανόμαστε τις συνέπειες της ε, θρησκευτικής ε, έντασης ε, και πρέπει να την μειώσουμε. Και νομίζω πως είπα αυτό το πνεύμα έχει γραφτεί το κείμενό μου. Δεν είναι κατά της Σαουδικής Αραβίας ούτε είναι κατά του Ιράν. Είναι υπέρ της ειρήνης και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να το ξαναδείτε. Για τον ρόλο του Ιράν στις άλλες συγκρεώσεις τώρα δεν θα ρωτήσω τη συνάδελφο αλλά δεν είναι τόσο απλό ότι κάθε κάποιο το χεράνει και δίνει διαταγές στην Ιεμένη π.χ. δεν ξέρω πόση επιρροή έχουν στο Λίβανο θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σε μια πολιτική λύση που σαφώς υπάρχει μεγάλος ε, ρόλος ε, σε σχέση με τη Συρία, αλλά και στην καταπολέμηση του Ντάις. Δηλαδή σε κάθε χώρα υπάρχουν διαφορετικές επιρροές και πρέπει να το συζητήσουμε εκτός της συνεδρίασης ε, προς την κυρία Σάκη, που ξέρω ότι ενδιαφέρεται σοβαρά για τα ζητήματα. Κοιτάξτε. Ναι, είχαν, κάνανε εκλογές και έχω ακούσει τα όσα έχουν υποθεί για την ποιότητα των εκλογών. Ναι, συγγνώμη, θέλω να κοιτάω και τους συναδέλφους. Ε, είμαι παλαιών αρχών. Για την ε, ημερομηνία των ε, εκλογών ίσως καθυστέρησε λίγο την πρόοδο, αλλά δεν ξαναγράφεται εδώ πέρα η πυρηνική, η, η πυρηνική συμφωνία. Είχαμε ψήφισμα την στιγμή της ε, συμφωνίας όταν είχε έρθει η κυρία Μογκερίνη. Οπότε πρόκειται για μια πιο μακροπρόθεσμη έκθεση και προσέγγιση. Ναι, τελειώνω. Μεταρρυθμιστές τώρα σε σχέση με τους πιο σκληροπυρηνικούς ε, πρέπει να το δούμε ρεαλιστικά. Λοιπόν, καλώς ορίζω τις ε, προτάσεις που έγιναν από τους συναδέλφους. Ο κύριος ε, Σάριος Βόλσκι μίλησε για αντικατοπτρισμούς. Θα το κρίνουμε. Δεν νομίζω να είναι αντικατοπτρισμός. Νομίζω πως υπάρχει μια στιγμή, ένα παράθυρο ευκαιρίας. Και τελειώνω. Όταν ο κύριος Κίλαμ είπε ότι πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις δηλαδή πυρηνική συμφωνία και τα ανθρώπινα δικαιώματα πριν από τίποτε άλλο. Διαφωνώ εδώ πέρα και νομίζω πως έχουμε τις συζητήσεις στις πολιτικές μας ομάδες, αλλά πρέπει να δούμε τις τροπολογίες και να διατηρήσουμε το γενικότερο ύφο. Τον Ιούλιο είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Περνάμε στο σημείο 7. Έχουμε τώρα την ευκαιρία να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων για την 20η ε, επέτειο από τη σύναψη της συνθήκης για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών, μια σημαντική ημερομηνία. ...164 χώρες έχουν ε, κυρώσει τη συνθήκη. Τελευταία ήταν η Αγγόλα νομίζω. Και 80, σε 85 χώρες λαμβάνουν χώρα επιθεωρήσεις αλλά βλέπουμε ότι η Βόρεια Κορέα συνεχίζει να κάνει δοκιμές και η συνθήκη παρά τις τόσες υπογραφές έχει την αδυναμία ότι δεν την τήρουν όλοι και έχουμε δυσκολίες ε, αλλά αυτό αφορά γενικότερα τις ε, σχέσεις ε, της διεθνής ότι είμαστε πάλι σε μια δύσκολη κατάσταση. Φεντερίκα, τώρα συζητήσαμε και το Ιράν και σε ευχαριστούμε και πάλι για την συμφωνία που πετύχατε και ελπίζω έτσι να περιοριστεί λίγο ο αυτοματισμός αυτός της απόκτησης πυρηνικών όπλων. Νομίζω λοιπόν πως είναι μια πολύ σημαντική δουλειά αυτή. και πρέπει να θυμόμαστε την συμφωνία και να είμαστε κάπως πιο ενεργοί. Και χαίρομαι ε, και για το ότι είναι αντιπρόεδρος εδώ πέρα σήμερα, αλλά και ο κ. Σέρμπο, ο οποίο είναι εκτελεστικός γραμματέας του οργανισμού, απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την δουλειά που κάνει. Μέχρι τις 10 ε, μπορούμε να μιλήσουμε γιατί μετά πρέπει να πάει στην Ολομέλεια η κυρία Μογκερίνη. Και θα δώσω μετά την Φεντερίκα τον λόγο στον κύριο Σέρμπο για να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων. Λοιπόν, έχετε τον λόγο. Uh, Ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι σήμερα εδώ με σας και ειδικά με τον δόκτορα Ζέρμπο. Είχαμε συνεργαστεί στην Βιέννη πριν από λίγες εβδομάδες ε, ορτάσαμε την 20η επέτειο της συνθήκης και τη δουλειά που έχουμε μπροστά μας τα επόμενα 20 χρόνια. έτσι ώστε η συνθήκη να λειτουργήσει ως το δυνατόν καλύτερα. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας, κύριε Πρόεδρε, για την συνεδρίαση αυτή. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η συζήτηση στην ΑΦΕΤ. Ο ρόλος των κοινοβουλίων είναι ένας ρόλος κλειδί και νομίζω πως είναι ήδη ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αγαπητό μου φίλο γιατί έχει εργαστεί στον τομέα της συνθήκης με ενέργεια και αφοσίωση πραγματικά αξιοθαύμαστη. Και πρέπει να πω πως ε, συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά. Και πρέπει να πω πως πριν αναλάβω αυτήν την θέση ε, τον ε, γνώριζα και νομίζω πως ο οργανισμός έχει κερδίσει από την εργασία του. Η συνθήκη είναι πολύ αποτελεσματική συνθήκη. Μετά 20 χρόνια από την υπογραφή της, οι πυρηνικές δοκιμές είναι πλέον μια ανομαλία. Ε, δεν έχουν σταματήσει όπως είπατε, αλλά είναι κάτι το τελείως ε, ασυνήθιστο και βεβαίως διεξάγονται ενάντια θέληση της ε, διεθνούς κοινότητας. Υπάρχει λοιπόν μια συνένεση, μεγάλη διεθνής συνένεση, για την συνθήκη και ο οργανισμός της συνθήκης είναι επίσης αποτελεσματικός παρά το ότι εξακολουθεί να είναι ακόμα προσωρινός είναι παγκόσμιος στην παρουσία του και κάνει κάτι που δεν μπορεί να κάνει καμία χώρα μόνη της δηλαδή συλλέγει και αναλύει δεδομένα από ολόκληρο τον κόσμο με την επιστημονική εμπλοκή που είναι εντυπωσιακή πραγματικά και με συνεισφορά από πολύ διαφορετικές χώρες. Έχει το δίκτυο ολοκληρωθεί κατά 85% και εδώ πέρα θα ήθελα και πάλι να συγχαρώ τον δόκτωρα Ζέρμπο και την ομάδα του για την εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει. Θα ήθελα να υπογραμμίσω την σημασία της διεθνούς τεχνικής συνεργασίας. Οι δικοί από χώρε ε, τόσο διαφορετικές όπως το Ιράν και το Ισραήλ ή η Ρωσία και οι Ηνωμένε Πολιτείες συνεργάζονται στην συλλογική αυτή προσπάθεια και κάθε ε, κράτος μέλος συνθήκης ε, εποφελείται από το έργο αυτό, από τις τεχνικές εργασίες και θα ήθελα να πω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη μας όλα έχουν παίξει σημαντικό ρόλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και θα συνεχίσει να είναι ο βασικός θα έλεγα υποστηρικτής του έργου και του οργανισμού. Και τα 28 κρατημέλη έχουν κυρώσει τη συνθήκη. Τακτικά ερχόμαστε σε επαφή με τις ε, χώρες του παραρτήματος 2 που δεν έχουν ακόμα κυρώσει ε, ή υπογράψει και κάνουμε αυτές τις επαφές ε, συντονισμένα και 28 χώρες ε, για να γίνει πραγματικά παγκόσμια η συνθήκη και παρέχουμε και σοβαρή χρηματοδότηση στον οργανισμό πάνω από 18 18,5 εκατομμύρια ευρώ. Και παρέχουμε και βεβαίως ε, τεχνική αρρωγή, εμπειρία στη γραμματεία κτλ. Ανέφερα λοιπόν τις επαφές με τις χώρες του παραρτήματος 2 Ξέρετε πόσα αυτά χρειάζονται για να γίνει παγκόσμια η συνθήκη και να τεθεί ενισχύ. Εμείς συνεργαζόμαστε ιδιαίτερα με αυτές τις χώρες με τρόπο συντονισμένο και με άλλους εταίρους και με τη στήριξη του οργανισμού και ασχολούμαστε ιδιαίτερα με τις ανησυχίες ασφαλείας των χωρών, ασχολούμαστε με περιφερειακά ζητήματα τονίζουμε τα ωφέλη και στον τομέα των πολιτικό και στον τομέα της ασφάλειας και φροντίζουμε βεβαίως να, υπάρχει, να υπάρχουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή της συνθήκης, κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους Αμερικανούς φίλους μας. Για τις χώρες του παρατήματος 2 θα ήθελα να αναφέρω τον ιδιαίτερο ρόλο των κοινοβουλίων. Επειδή και εγώ ήμουν η ίδια βουλευτής, γνωρίζω πάρα πολύ καλά πως η επαφή με εθνικούς βουλευτές είναι πολύ σημαντική, γιατί σε τελική ανάλυση η απόφαση για κύρωση βεβαίω επαφείται στα κοινοβούλια, σε δημοκρατικές χώρες τουλάχιστον, και οπότε η επαφή με τους συναδέλφους στα εθνικά κοινοβούλια ή σε διακοινοβουλευτικά φόρα είναι πάρα πολύ σημαντική για να δημιουργηθεί απαραίτητη συνένεση. προφανώς επαφίεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καθορίσει τους καλύτερους τρόπους ε, προόδου, μπορεί να είναι ένα ψήφισμα ή δικτύωση, πώς θα μπορέσουμε να δικτυωθούμε καλύτερα σε διακοινοβουλευτικές διασκέψεις, συντονισμός ε, και το πώς θα ενθαρρύνουμε επαφές ε, ευρωβουλευτών με εθνικούς βουλευτές, ειδικά των χωρών του παραρτήματος 2. Και είμαι σίγουρη πως ο οργανισμός της συνθήκης ε, είναι διατεθειμένος να βοηθήσει το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιστεύω πραγματικά πως έχουμε την αξιοπιστία, έχουμε τα μέσα και τις ε, ικανότητες ε, και την ποικιλομορφία για να έρθουμε σε επαφή με πολλές χώρες ανά τον κόσμο. Επίσης να αναφέρω ότι έχουμε την ικανότητα να συνεργαστούμε με την κοινωνία των πολιτών, τις ΜΚΟ και με δίκτυα βουλευτών μεταξύ των οποίων ε, το PNND, το δίκτυο βουλευτών για, την, ε, για τον πυρηνικό αφοβλισμό Τέλος, περιφερειακή διάσταση. Εδώ πέρα μπαίνουμε στην πτυχή που είναι πιο ενδιαφέρουσα από γεωπολιτική σκοπιά. Προσωπικά Είμαι πεπισμένη ότι η ταυτόχρονη κύρωση από κάποιες χώρες θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική ε, προοπτική συνεργασία σε κάποιες ε, περιοχές. Υπήρχε μια ταυτόχρονη υπογραφή από την Ινδία και το Πακιστάν. Θα έστελνα ένα ισχυρό μήνυμα που θα πήγαινε πέρα από το θέμα των περιπολικών ή από την Αίγυπτο και το Ισραήλ θα μπορούσε να αποτελέσει την βάση ε, για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης αλλά και για μια ζώνη η οποία θα είναι ελεύθερη από πυρηνικές δοκιμές που είναι ένα πρώτο βήμα για να είναι ελεύθερη και από όπλα μαζικής καταστροφής. Στο διεθνές πλαίσιο που έχουμε συμφωνήσει. Προφανώς πρόκειται για έναν κύκλο λοιπόν ε, ή δεν ξέρω ε, το αυγό και η κότα. Μπορούμε να περιμένουμε την περιφερειακή διάσταση για να γίνουν τέτοια βήματα ή το αντίστροφο, να γίνουν τέτοια βήματα για να υπάρξουν περιφερειακές εξελίξεις. Κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε και είμαι σίγουρη πως υπάρχει εδώ πέρα περιθώριο μιας προσέγγισης που θα είναι αμοιβαία υποφελής. Θα σταματήσω εδώ λοιπόν και θα δώσω τον λόγο στον αγαπητό μου φίλο για να μας πει πιο λεπτομερώς το τι κάνει κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ όλους και εκείνον που μας δίνει την ευκαιρία να εορτάσουμε την 20η επέτειο με τρόπο ουσιαστικό. Σας ευχαριστώ πολύ για την κοινοβουλευτική διάσταση της αρχής Σεπτεμβρίου έχουμε το IPC με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και εκεί μπορούμε θα μπορούσαμε να θέσουμε το θέμα αυτό. Να το συζητήσουμε με τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Μογκερίνη. Ευχαριστώ και τους ε, αγαπητούς και αξιότιμους ευρωβουλευτές που μας ε, κάλεσαν εδώ για να μιλήσουμε για την ε, συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ την κυρία Μογκερινή, η οποία είναι καλή φίλη και όπως είπε, συναντηθήκαμε σε ό,τι αφορά το πλαίσιο των κοινοβουλευτικών σχέσεων και ξεκίνησε αυτή η διαδικασία πριν από τρία χρόνια. Και βρισκόμαστε λοιπόν εδώ σήμερα. Κυρία Μογκερίνη, νομίζω ότι επέδειξε η κυρία Μογκερίνη μεγάλη ηγεσία, γιατί έφερε το θέμα αυτό στα υψηλότερα κλιμάκια. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να το προβάλλουμε το θέμα αυτό, γιατί στην πράξη δεν είναι πολλοί αυτοί που μιλάνε για την ε, συνθήκη αυτή, για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών, αλλά η Ευρώπη μιλάει για το θέμα αυτό, γιατί αντιπροσωπεύει και το 40% του προπολογισμού τη οργάνωση αυτή. Και έτσι αναπτύξαμε ένα διεθνή σύστημα εποπτείας και κινούμαστε προς την ολοκλήρωση ενός καθεστώτος επαλήθευσης, μεταξύ άλλων και χάρη στην ε, χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν είναι ευθύνη μας να σας ενημερώνουμε για το τι έχουμε πετύχει με τη δική σας ε, χρηματική και πολιτική υποστήριξη και πώς με την ηγεσία σας μπορούμε να πετύχουμε ε, πράγματα πολύ σημαντικά για τη διεθνή ασφάλεια και η ειρήνη χάρηκα που άκουσα στη συζήτησή σας και για το Ιράν και από εκεί θα ξεκινήσω. Ήταν ενδιαφέρον το ότι σας άκουσα αξιότιμοι ευρωβουλευτές να μιλάτε για το Ιράν. Το πώς προσεγγίζετε και πώς σκοπεύετε να προχωρήσετε το θέμα αυτό. Να πω το εξή. Η κυρία Μογκερίνη υποστηρίζει ε, το πώς θα μπορούσε να ενταχθεί το CPTPP στην συνθήκη με το Ιράν, στη συμφωνία με το Ιράν. Και υπήρξε μία χαμένη ευκαιρία, αν και θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι εγώ είμαι μερελεπτικός και πάντα θα μιλήσω για θέματα της συνθήκης αυτής. Αλλά θεωρώ ότι σε ό,τι αφορά τη σύναψη της συμφωνίας αυτής υπάρχει τρόπος να πείσουμε τους Ιρανούς να εξετάσουν την επικύρωση της συνθήκη για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών, γιατί πιστεύουμε ότι το θέμα αυτό είναι, αν θέλετε, και λίγο ε, ένα θέμα το οποίο έχει καθιερωθεί έτσι. Και το Ιράν έχει επιδείξει καλή θέληση Μας έχουν μιλήσει για παράδειγμα για μια βαθμία προσέγγιση για το θέμα αυτό και εφαρμόζοντας και υλοποιώντα τη συμφωνία με το Ιράν, θεωρώ ότι υπάρχει μια ευκαιρία για εσά, τους Ευρωβουλευτές σταδιακά να εισαγάγετε ε, το θέμα τη ε, ένταξης της συνθήκης στη συμφωνία αυτή για να επαναληφθούν και όσα ξεκίνησαν πριν από κάποιου μήνε για να επανέλθει το Ιράν στα διεθνή φόρα. Εδώ λοιπόν αυτό αποτελεί μια χαμένη ευκαιρία. Και μυρίσαμε και για την Συρία. Άλλη χαμένη ευκαιρία. Όντω, η επικυρίωση τη Συρία δεν είναι προαπαιτούμενο για να τεθεί σε ισχύ η συνθήκη αυτή, αλλά για να οικοδομηθεί μια σχέση εμπιστοσύνη. Αν η Συρία μπει στη συνθήκη για τα χημικά όπλα, θεωρώ ότι η συνθήκη αυτή ήταν σημαντική. Θα είχε ληφθεί υπόψη από τον πρόεδρο Ασάντ. Το έχει εξετάσει το θέμα της υπογραφής και της επικύρωσης της συνθήκης. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή υπάρχουν ε, χαμένες ευκαιρίες, γι' αυτό λοιπόν ζητούμε από εσάς, τους Ευρωβουλευτές, και από την κυρία Μογερίνη να αναλάβετε την ηγεσία του θέματος, να προσεγγίσετε και τη ΣΥΠΑ, γιατί ο πρόεδρος Ομπάμα κατέστησε σαφές ότι ήταν πρόθεσή του 2009 ήδη να περάσει το CTBC, CTBT ε, προσωπική ρωσία από τη Γερουσία, αλλά πολύ απλά δεν έχει ε, Του αριθμού, τα αριθμητικά στοιχεία που χρειάζονται, την υποστήριξη που χρειάζεται. Αυτό έχει να κάνει και με τη δημοκρατία. Εκεί λοιπόν έχουν τα πράγματα και εδώ έχουν κολλήσει μέχρι και σήμερα. Πολλά λοιπόν θα πρέπει να γίνουν από δική σα πλευρά. Όπω ε, είπε και η κυρία Μογκερίνη και ο κύριο Πρόεδρο, πολλά μπορούμε να κάνουμε για να μπει το θέμα αυτό στη συζήτηση, γιατί η συζήτηση για την επικύρωση τη συνθήκη είναι στα δικά σα χέρια και υπάρχει ευκαιρία να συνομιλήσετε και με τους ομολόγους σας. Γι' αυτό λοιπόν από εσάς ζητάμε να μας βοηθήσετε από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν, μπορούμε, δεν μπορείτε ε, να πληρώνετε κατά 40% τα θέματα αυτά και μετά να ε, επιτρέπετε να συνεχίζονται αυτές οι τριβές τα τελευταία 20 χρόνια. Πριν από 10 ημέρες συναντήθηκα με διάφορους ε, πολιτικούς ηγέτες, με, μίλησα και με τον Πρωθυπουργό Νετανιάου για να μιλήσουμε την εφαρμογή, για την εφαρμογή της συνθήκης αυτής. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ήταν μεγάλη τιμή για μένα και νομίζω ότι δείξαμε πολλά θέματα. Από τα περιφερειακά ζητήματα κοιτάξαμε το τι επιδιώκει και στο διεθνές προσκήνιο το Ισραήλ. Ο Πρωθυπουργός Νετανιά, όπω ξέρετε, ε, προγραμματίζει, ε, επισκέπτεται μάλλον την Ανατολική αλλά και την Βετρική Αφρική. Και ένα από τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν ήταν Πώς μπορούμε να συγκεντρώσουμε μία θετική διάθεση προς το Ισραήλ και σε ό,τι αφορά τα όσα κάνει για την περιφέρεια αυτή. Ένα θέμα λοιπόν είναι και αυτή η συνθήκη για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών. Δεν έχουν να χάσουν άλλωστε τίποτα, μόνο να κερδίσουν μπορούν. Υποστήριξη προς το Ισραήλ δηλαδή και προς το ρόλο του Ισραήλ στην περιοχή και για το θέμα της Παλαιστίνης, το οποίο ακούσατε κάποιοι από εσά σήμερα. Καλούμε να επικρατήσει η λύση των δύο κρατών. Αυτό υποστηρίζει και τη διεθνή κοινότητα. Θα μπορούσε λοιπόν να χρησιμοποιηθεί ως μόχλευση αυτή η συνθήκη. Να πω το εξής, ότι με τα δικά σας χρήματα, με το δικού σας πόρους έχουμε πετύχει πολλά και στην διεθνή κοινότητα πλέον θα παρέχουμε όχι μόνο ένα διεθνές ε, σύστημα ελέγχου και εποπτείας, το οποίο κάποιοι θα αποκαλούσαν μια, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ε, σύγχρονης διεθνούς κοινωνίας. Και αυτό το παρέχουμε στην διεθνή κοινότητα, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα επικυρωθεί η συνθήκη. Και αυτό με φέρνει στη Βόρεια Κορέα. Είναι ένα θέμα η Βόρειος Κορέα. Είμαι απογοητευμένος, επιτρέψτε μου να πω. Γιατί σε ό,τι αφορά τη Βόρειο Κορέα δεν κάνει κανείς ε, καν τη σύνδεση με τη συνθήκη. Γιατί το μορατόριο ε, για τη χρήση των πρινικών θα αποτελούσε ένα τεράστιο επιτεύγμα ένα τεράστιο ορόσημο για την επίλυση του ζητήματος στην χερσόνησο της Κορέας. Δεν αναφέρεται καν η συνθήκη όταν μιλάμε για την επίλυση του ζητήματος της Κορέας. Και εδώ πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να ασκήσει επικοδομητική πίεση, γιατί είναι δική σας η χρηματοδότηση. 40% των πόρων προέρχονται από εσάς. Θα πρέπει να προασπιστείτε λοιπόν τους σπόρους αυτούς και να επιδιώξετε να υπάρξει μεγαλύτερος αντικτύπος. Μπορώ να μακρηγορήσω πολύ, αλλά νομίζω ότι πιο σωστό και ορθό θα ήταν να σας αφήσω εσάς να θέσετε ερωτήσεις, γιατί μίλησε για το Διεθνές Σύστημα Επιτήρησης και Εποπτείας η κυρία Μογκερίνη και επαναλαμβάνω ότι χρειαζόμαστε τη δική σα ηγεσία για να υπάρξει επικύρωση τη συνθήκη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και σα ευχαριστώ που βρίσκουμε εδώ σήμερα. Εμεί σα ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ε, σας ευχαριστώ, λέει ο κύριος Φραν. Να σα μιλήσω εκ τη της ε, Αυστρίας, της χώρας που φιλοξενεί τον Οργανισμό Ενεφορμή της Συνθήκης. Ε, στην Βιέννη και πάντοτε ξέρετε ότι τιμούμε τις να Μας αρέσουν. Δηλητηριάζουν το περιβάλλον ε, οι ποινικές δοκιμές, αλλά και το πολιτικό περιβάλλον, γιατί οδηγεί σε φόβο, δυσπιστία, απομόνωση και έχουμε ε, δει ότι όσοι κυβερνήσεις για όλα αυτά τα εργαλεία θανάτου έχουν πάρα πολλά λεφτά. Όμως είπαμε όσοι έχουμε επισκεφθεί και τη με το Ναγκασάκι ε, ποτέ δεν έχουμε γυρίσει στο σπίτι ακριβώς όπως ε, φύγαμε και βέβαια η συνθήκη ακόμα δεν έχει τεθεί σε ισχύ σε πάρα πολλές χώρες οπότε από εμά εξαρτάται και όχι μόνο βέβαια από εμά να συντοπίσει όλος ο κόσμος την ε, σημασία του πράγματος είναι σημαντικό αλλά βέβαια Έχουμε την Προπαρασκευαστική Επιτροπή, η οποία θέλει να προστατεύσει τον κόσμο και όσον αφορά τα αποτελέσματα των ε, φυσικών καταστροφών. Α πούμε, στην Φουκουσίμα, όταν το εργοστάσιο καταστράφηκε, τότε το διεθνέ σύστημα βοήθησε την κυβέρνηση τη Ιαπωνία. Επίση, είναι πάρα πολύ σημαντικό, μην ξεχνούμε ότι έχουμε διάφορα ηλεκτρονικά τα οποία καταγράφουν ε, οτιδήποτε γίνεται στον φλοιό της γης και χτυπάει σαν γερμός όταν υπάρχει ένα θέμα όταν ε, γίνει κάτι το που βγίζει σε τσουνάμι. Οπότε οποιοδήποτε δεν προσυπογράφει και δεν προσχωρεί στη συνθήκη, τότε αυτό το οποίο κάνει είναι να απαρνείται, να απεμπορεί τι ε, ευθύνε του σαν μέρο τη διεθνού κοινότητα. Οπότε και εγώ ταπεινά έχω να σα προτείνω ότι ίσω είναι χρήσιμο να γίνει μια συζήτηση στην Ολομέλεια για αυτό το θέμα κατά την 20η επέτειο. Οπότε και εμείς έτσι θα δείξουμε ότι υποστηρίζουμε την ε, δουλειά σας. Ευχαριστώ. Ε. Ο επόμενος. Συγγνώμη, καθυστέρει λίγο η διερμηνία, γι' αυτό δεν αντιδρώ αμέσως. Μία ερώτηση έχω μόνο εγώ. Πώς μπορούμε να δούμε τις εμπορικές σχέσεις ε, και να τις χρησιμοποιήσουμε για να πιέσουμε για μη διάδοση. συγκεκριμένα για Ινδία, Πακιστάν και Αίγυπτο και Ισραήλ. Για Κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Θυμάστε τις συζητήσεις στην τελευταία συνεδρίαση και στην τελευταία διάσκεψη για τη μη τη συνθήκη της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων. Ξανά η ερώτηση, λοιπόν. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ρήτρε στις εμπορικές συμφωνίες για να προωθήσουμε την συνθήκη. κύριος Καν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καλώς όρισαν οι καλεσμένοι μας. Πριν γίνω ευρωβουλευτής ήμουνα αντιπρόθεσης οργάνωσης ε, για την ειρήνη του των δημάρχων. Οπότε επισκέφθηκα τότε Ναγκασάκια και Χειροσύμα και είδα την Φρίκη που επικρατεί εκεί για όσα έγιναν. Ναι, είναι τρομερό να μην προσυπογράφουν κάποιες χώρε. Αλλά για πετε μας, τι άλλο μπορεί να γίνει. Πώς το ευρωπαϊκό μπορεί να σα βοηθήσει κι άλλο στο έργο σα. Ξέρετε, έχω ειδική καταγωγή. Και βέβαια ξέρουμε τι γίνεται από πλευρά πυρηνικών στην Ινδία και Πακιστάν. Τι λένε αυτοί που ξέρουν. Πάντως, στη δεκαετία 90 και στην Μέση Ανατολία κατεβληθεί προσπάθεια, ούτως ώστε εκεί να μην αναπτυχθούν πυρηνικά. Και κάναμε ό,τι μπορούσαμε, έχουμε και την συμφωνία με το Ιράν, αλλά έχουμε και το Ισραήλ, γιατί πολλοί θεωρούν λοιπόν υπάρχουν εκεί πέρα περί τις 200 ε, πυρηνικές βόμβες. Για πετε μας εσείς στο όλο αυτό το τοπίο αυτά πώς συντεριάζουν. Ο πρόεδρος εκτός μικροφώνου δίνει σε κάποιον το λόγο. Αν ε, κύριε Μογκερίνη. Σε σχέση με το πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα και τι συμφωνίες συμφωνίε, ώστε να ασκήσουμε πίεση, αν ρίξετε μια βαθιά ε, τι γίνεται στο δεύτερο παράρτημα στις σχετικές χώρες. Ε, ναι, αυτό έχει απασχολήσει επανειλημμένα και το Κοινοβούλιο Κίνα, Ιράν, Βόρεια Κορία, Ινδία, Πακιστάν, Αίγυπτο και Ισραήλ. Γιατί για όλε αυτέ τι χώρε σχεδόν για όλες αυτές, έχουμε ασκήσει τέτοιου είδου πίεση. Οπότε βέβαια και είναι θέμα πολιτική επιλογή Μέχρι ποιο βαθμό θα χρησιμοποιήσει κανεί αυτά τα μέσα. Ε, Όποτε θέλετε να το συζητήσουμε. Αλλά βέβαια γνωρίζω ότι είναι θέματα αυτά οικονομικά, είναι θέματα εμπορικά, αλλά και γεωπολιτικά. Πέραν από το πάντως, οπότε θέλετε να το συζητήσουμε εδώ στο Κοινοβουλίο και στην Ολομέλεια. Βέβαια, χτες το απόγευμα είχαμε στην Ολομέλεια πολύ λίγο λιγότερους βουλευτές από ό,τι σήμερα εδώ στην Άφετ Γι' αυτό και με ενδιαφέρει τόσο πολύ να έρχομαι στις κοινοβουλευτικέ επιτροπές. Εντάξει, δεν λέω ότι μου αρέσει και το ημικύκλιο, τέλος πάντων. Πάντω σα τονίζω το εξή. όπως αναφέρατε ότι η υπόθεση αυτή της συνθήκης και του οργανισμού για τη συνθήκη είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το υποστηρίζει η Ένωση και οικονομικά, σημαντική οικονομική βοήθεια δίνει και αυτό γιατί είναι κάθε αυτό σημαντικό, αλλά είναι και σημαντικό γενικότερα για το θεματολογιό μας. Για την μη διάδοση, για τον αφοπλισμό, για τα πυρηνικά, για την ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό θέμα για την ε, πολιτική ασφάλεια. Επίσης, αυτό έχει σχέση και με το θεματολόγιο μας για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια συνεργασία στα περιφερειακά συστήματα σε όλο τον κόσμο αυτό. Ακόμα, ακόμα δεν έχει επιτευχθεί. Άρα, με τη δουλειά που γίνεται για αυτή τη συνθήκη, μπορούμε να βάλουμε το λιθαράκι μας για διάφορες περιοχές του κόσμου, όπως αναφέρετε και εσείς, για το Παγιστάν ή και για τη Ανατολή, Φερρυπίνου. Νομίζω ότι αξίζει η προσπάθεια που καταβάλλετε. Είναι πολύτιμο το έργο σας. Έχει ευρύτερη σημασία πολιτικά και αξία. Για την ειρήνη στον κόσμο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μας μίλησε κύριε για το η κυρία Μογγερίνη. Να, αυτή είναι η επικοδομητική πίεση. Ξέρετε, προέρχομαι την Πουρκίνα Φάσο και το εμπόριο είναι πολύ σημαντικό. Και μπορώ να διαπιστώσω πόση πίεση αποδίδει. Να, ένα μικρό παράδειγμα. Όταν επισκεπτούμε χώρε όπω την Αγγόλα, όπως ε, ανέφερε ο πρόεδρο, είναι τι τελευταίε χώρε που προσεχώρησαν ε, στην συνθήκη. Όταν λοιπόν κανεί ε, συνεννοείται με χώρε, χώρε, όταν συζητάμε για μια μη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλεία, βεβαίω και υπάρχει επικοδομητική πίεση. Έχετε υπογράψει τη συνθήκη, έχετε κυρώσει το πρωτόκολλο, έχετε κάνει το α, το β, το γ, όταν παζαρεύεται η θέση αυτή στο Συμβούλιο Ασφαλεία. Να, πόσο ωφελεί για χώρες από την Αγγόλα αυτή η πίεση και πολλές που χώρες ώστε να μπορούν να μπουν στα διεθνή φόρα. Θα πρέπει να αποδείξουν ότι το αξίζουν. Πρέπει, πρέπει να ασκείται τέτοιου είδους πίεση. Τώρα, για αυτό που τώρα είναι υποσυζήτηση. Η Ινδία δηλαδή να προσχωρήσει στην ε, ομάδα για τα πυρηνικά. Θέλετε γιατί δεν ε, αναφέρεται τη συνθήκη. Είναι βέβαια για Ινδία και Πακιστάν που θέλουν να μπουν σε αυτή την ομάδα για τα παιχνικά το Suppliers Group. το, για να το πούμε, εντάξει, δεν, δεν είναι τίποτα αλλά αυτό που κάνουμε είναι ότι κάνει ο ψαράς. Όταν τα ψάρια φαγώνονται μεταξύ τους, τότε το εκμεταλλεύεται ο ψάρας. Οπότε έτσι και εμείς σιγά σιγά περιμένουμε για να δούμε το πώς θα καταφέρουμε και εκεί να ισχύσει η συνθήκη. Οπότε όπως η Ινδία και Πακιστάν έτσι θέλουμε και η Αίγυπτος, το Ιράν και το Ισραήλ να προχωρήσουν στη φάση που είπε η κυρία Μογκερίνη. αυτήν την κοινή κύρωση τη συνθήκη. Κάποιοι λένε ότι αυτό είναι αδύνατο. Μα τίποτα δεν είναι αδύνατο. Μα ε, τα έχετε καταφέρει στα πλαίσια του Ιράν. Ε, πήρε χρόνο, αλλά το καταφέρατε με το Ιράν. Το είπατε κύριε Μαγερίνη. Και νομίζω ότι αυτό και θα πρέπει να κάνουμε. Αλλά λέμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε για αυτή τη συνθήκη απαγόρευση των δοκιμών. Ε, το, το κάνατε για το Ιράν. Είναι σκληρό να κάνει στον κόσμο να. Ε, και δύσκολο να κάνει στον κόσμο να κάθεται στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Αλλά αυτό μπορεί να αποδώσει. Και μετά κανεί είναι ευτυχή για αυτό που καταφέρει. Ε, μετά από μια εικοσαετία α κάνουμε κάτι. Α κάτσουμε γύρω από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ας είμαστε ρεαλιστές γιατί είναι δύσκολη η πραγματικότητα σκληρή. Είναι δυνατόν να επενδύουμε τόσα πολλά σε ένα θέμα όπως η μπορούμε των δοκιμών και μετά να το εγκαταλείπουμε ούτως ώστε να λέει ο κόσμος ότι να ξέφτησε η συνθήκη. Γιατί να συνεχίσουμε να δίνουμε λεφτά για κάτι αφού δεν υπάρχει φως στην άκρη Να, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει να υπάρχουν ε, συζητήσεις και πάρα πολλοί βουλευτέ είπαν ότι θα πρέπει το θέμα αυτό να κατέβει στην Ολομέλεια. Το είπε και η κυρία Μογγερίνη ότι εδώ έχουμε περισσότερου βουλευτές από ό,τι έχουμε στην ε, Ολομέλεια, στο ημικύκλιο. Εντάξει, ξέρω ότι είναι ανώτερο όργανο, αλλά όταν εκεί έρχονται αυτά τα θέματα, ε, τότε φαίνεται προς όλο τον κόσμο το πόσο σημαντική είναι κάποια υπόθεση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτό θέλουμε να μείνει το θέμα στο επίκεντρο της επικαιρότητα. Οπότε πρέπει να σας ευχαριστήσω θερμότατα για το πόσο μας έχετε στηρίξει που μας καλέσατε σήμερα μαζί με την υπατή εκπρόσωπο. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε αυτό το θέμα να εξεφτίζει. και κυρίως ε, σε σχέση με αυτούς που βοηθούν τόσο οικονομικά. Αν έχω λόγια σας ευχαριστήσω να, και στο ΝΑΤΟ μπορεί κάτι να γίνει. Έχουμε την διάσκεψη της ε, Λιουμπλιάνα και είχα πάει εκεί και είχα μιλήσει για τη συνθήκη. Και πάρα πολύ στο ΝΑΤΟ. Δεν είχαν καν ακούσει επί πάρα πολύ καιρό για τη συνθήκη πόλευσης δοκιμών. Άρα να, και σε κείμενα του ΝΑΤΟ να την αναφέρουμε την ε, συνθήκη. Έχουμε εκεί τρόπο παντού χώρε της που συμμετέχουν. Επομένω να συνεχιστεί στι 8 εναπομείνωσες χώρε. αυτή η πίεση γιατί μετά από μια εικοσαετία, ετία τώρα μπορούμε να δούμε προσέγγιση στον στόχο την εφαρμογή τη συνθήκη. Πολύ σημαντικό, γιατί τόσο καιρό περιμένουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο. Μόνο όλη αυτή η διαδρομή και αυτή είναι κομμάτι αυτή τη ευκαιρία, τη ευκαιρία τη διαδρομής και έτσι ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε στο στόχο μα. θα τον πετύχουμε το δυνατή σχέση συνθήκη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε οπωσδήποτε και την στήριξή μας, αν την χρειάζεστε. Νομίζω πως θα τα ξανασυζητήσουμε αυτά τα ζητήματα και με τους συναδελφούς στα Εθνικά Κοινοβούλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν και καλή επιτυχία στη δουλειά σας. Έχουμε και άλλο σημείο στην ερήσια διάταξη, μην φύγετε. Έχουμε άλλο ένα θέμα στην ερήσια διάταξη. Το είπα και πριν. Έχουμε το ζεύγος Γιουνούς από το Αζερβαϊτζάν και την γενναία κόρη τους που μας βασάνιζε εδώ πέρα να κάνουμε κάτι. Τα κατάφερε όμως. και ε, έτσι είναι οι κόρες με τους γονείς. Και ελπίζω να έχουν την ευκαιρία να μας πούν δύο λόγια για την κατάσταση στη χώρα τους για να συνεχίσουμε μετά τις 10. beginnen wir. Vielleicht sollen wir dann mit Herrn Yunus beginnen. Ε, μα, θα ξεκινήσουμε, τι θα μαζευτήκατε εκεί πέρα οι γυναίκες. So, λόγο έχει η κυρία Γιουνούς. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ ε, δύσκολα μετά τη φυλακή να πάρω το λόγο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω λίγο άγχος και θα σας παρακαλέσω να με συγχωρέσετε. <laughs> no, you cannot imagine the prison in... Όχι, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο έχει φυλακή στο Αζερβαϊτζάν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να πω, όπως είπα και στην κυρία Μοκερίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, μεγάλη υποστήριξη. Προς εμένα, προς τον ε, άντρα μου τον Αρίφ, ε, να ευχαριστήσω και για την υποστήριξη προς όλους τους φίλους και συναδέλφους που ε, φυλακίστηκαν. Ήταν τεράστιε οι πιέσει που δεχτήκαμε στο Αζερβαϊτζάν. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πρόεδρο Σούλτ, τον κύριο Έλμαρ Μπλόκ, την κυρία Πύρη, την κυρία Λούνατσεκ. Πολλέ ευχαριστίε γιατί χωρίς τη δική σα υποστήριξη δεν θα ελπίζαμε καν ε, να, έχουμε, να είμαστε ελεύθεροι, να είμαστε μαζί με τις οικογένειές μας και κατά τη διάρκεια της δίκης ειλικρινά δεν πίστευα ότι θα μπορέσει να έρθει η στιγμή αυτή της ελευθερίας. Να σας εξηγήσω δύο λόγια για το πώς έχουν τα πράγματα σήμερα στο Αζερβαϊτζάν. Γιατί νομίζω ότι στην Ευρώπη δεν κατανοείται, πραγματικά δεν κατανοείται τι χώρες υπάρχουν στα νότια του Καυκάσου εμείς ξεκινήσαμε στη Σοβιετική εποχή τον ακτιβισμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Σοβιετική Ένωση είχε μεγάλες πολυεθνικές φυλακέ. Ξέρετε τα πώς έχουν τα πράγματα αυτά. Σε ό,τι αφορά το Αζερμπαϊτζάν τώρα, σήμερα είναι ένα μικρό κράτο. Σε ό,τι αφορά και τι ε, φυλακέ, είναι μικρέ και εθνικέ. Το Αζερβαϊτζάν σήμερα είναι μέλος του ΑΣΑ, που συμβουλευτή της Ευρώπης, έχει, της Ευρώπης, έχει καλή πολιτική γειτονία. Και ένας από τους συναδέλφους μας μας είπε ότι, κοιτάξτε, πώς μπορούμε να συγκρίνουμε το Σερβαϊτζάν με την Σοβιετική Ένωση. Δεν μιλώ όμως για την εποχή του Στάλιν. Μιλώ για την εποχή του Γκουρμπατσόφ. Τώρα όμω σιγά σιγά πάμε προ την Σταλινική εποχή. Ο σύζυγό μου, Αρίφ, ε, συνελήφθηκε για πρώτη φορά το 1976. Και αυτό και οι του φίλοι προσπάθησαν να δημιουργήσουν εναλλακτικέ οργανώσει. Αλλά η έρευνά του στη Σοβιετική Ένωση ε, και του είπαν ότι δεν μπορούσαν πριν από την ε, επέτειο για τα Οκτωβριανά να, να φυλακίσουν νεαρούς. Έκαναν έρευνες. Τώρα τον συνελήφθη το 2014 και φυλακίστηκε στο ίδιο μέρος στο ε, Υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας του ξαναβγάλαν αυτή την υπόθεση του 1976 και του είπαν ότι είσαστε εχθρός μας. Εχθρό μα από το 76 και παρακολουθούμε την κατάσταση έκτοτε. Τον βασάνισαν γιατί τον ε, είχαν βασανίσει και από τα 16 του και αντιμετωπίζει προβλήματα. Το Ινστιτούτο για την Δημοκρατία δημιουργήθηκε το 1994 ως μη κυβερνητική οργάνωση του Αζερβαϊτζάν και εκεί συνεχίσαμε τη δράση μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ένα από τα βασικά καθήκοντα ήταν να φτιάξουμε ένα κατάλογο πολιτικών κρατουμένων. Ο, πριν ενταχθεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης ε, το Αζερμπαϊτζάν, είχα 760 ονόματα στην λίστα των πολιτικών κρατουμένων μου και απαιτήσαμε το Αζερμπαϊτζάν όταν μαζί με την ε, Αρμενία και τη Γεωργία εντάχθηκαν στο Συμβούλιο της Ευρώπης να ανταπεξέλθουν να επικυρώσουν και να, από τις πολιτικές τους δεσμεύσεις. Και διορίστηκε και ειδικό ενταλμένο για θέματα πολιτικών κρατουμένων. Και υπάρχουν λοιπόν, ε, κάνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά αυτή. Και από το 760 σε δύο ε, χρόνια απελευθερωθήκαν πολλοί. Πλέον μόνο 17 κρατούνται. Το 2010. Ο Κρίστοφερ Στράσερ ήταν ειδικό διταλμένο σε ό,τι αφορά τα θέματα πολιτικών κρατουμένων. Και ο κατάλογο ε, μεγαλώνει και πάει. 300 περίπου περιλαμβάνονται πλέον. Δεν έλαβε καν θεώρηση να μεταδεί στον Πακού το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο ειδικό εντονταλμένος του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν πήρε βίζα για να πάει στον Πακού. Ε, συνεργαζόμαστε στενά με το γραφείο του κυρίου Στράσερ και του χορηγούμε ε, υλικό για κάθε πολιτικό κρατούμενο. Το 2013 τον Ιανουάριο, στην διάσκεψη, όταν, ε, στη Σύνοδο, όταν συζητήθηκε το θέμα των πολιτικών κρατουμένων ε, στο Αζερβαϊτζάν και το σχετικό ψήφισμα, δεν είχαμε αρκετές φωνές. Τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν τάχθηκαν ε, ηχηρά υπέρ του ψηφίσματος από τους πολιτικούς Ουσιαστικά τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης έδωσαν πράσινο φως για τις φρικαλαιότητες και τα κατασταλτικά μέτρα. Ο Ιρμαναμέντεφοφ, ε, και άλλοι ε, ηγέτες ε, της αντιπολίτευσης συνελήφθησαν και ξεκίνησαν τα κατασταλτικά μέτρα. Το Νοέμβριο του 2014 ξεκίνησαν αυτά. Όταν ε, προείδρευε στη σχετική επιτροπή το Αζερβαϊτζάν στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Και εμείς θα ανεχόμαστε αυτά. Αν εκ των προτέρων είχαν κατασταλεί αυτά τα φαινόμενα σε ό,τι αφορά την καταπίεση της αντιπολίτευσης, μέσα σε έξι μήνες συνελήφθησαν όλοι οι ακτιβιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δημοσιογράφοι. Αλλά ένα φίλος μου μου είπε ότι, κοιτάξτε, εσεί είστε ένοχοι γιατί έχετε τόσο μεγάλη εμπειρία και πρέπει να κατανοείτε αυτό. Θα πρέπει να ξέρετε πότε θα σας συλλάβουν. Να φύγετε από τη χώρα πριν σας συλλάβουν. εσεί είστε Τι την κόρη σας φέρετε στι κάτω χώρε. Ξέρετε όμω, το Ίδρυμά μας ήταν πάρα πολύ δημοφιλέ στο Αζερμπαϊτζάν και έλαβα πολλές επιστολές. Μπακού Λέιλα Γιούνου χωρίς διεύθυνση, τίποτα. Τα λάμβανα αυτά τα γράμματα. Καταλαβαίνετε πόσο γνωστοί είμαστε. Ε, χρειάζεται ο κόσμο την υποστήριξή μας. Απλά θέλω να σα εξηγήσω ότι δεν είναι μόνο οι ακτιβιστέ τη κοινωνία των πολιτών που έχουν και ασκούν πίεση στο Αζερβαϊτζάν και ο κανονικό κόσμο, ο απλό κόσμο. Δεν ζει σε καθεστώς ελευθερία στη χώρα αυτή. Το 2008 στο ίδρυμά μα μια οικογένεια από τη βόρεια, από τη βόρεια επαρχία της ζερμπαιτζαν δύο ε, αδελφές ετών 14 δεν θέλω να μακρηγορήσω. Αλλά ο επικεφαλής ε, της αστυνομίας ε, της επαρχίας αυτής οργάνωσε την κλοπή, την ε, απαγωγή των κοριτσιών αυτών για οργανώσεις trafficking. Φυλακίστηκε λοιπόν ε, κάποιοι παρατραχάμενοι και τελικά ο αστυνομικό ε, διοικητή παραμένει στη θέση του και συνεχίζει το τράφικινγκ. Χτε δημοσιεύτηκαν ε, πληροφορίε από το Υπουργείο Εξωτερικών τη Αμερική για θέματα διακινητών και η υπεύθυνοι και η ξέρετε που είναι, στα κλεμάκια του Υπουργείου Δικαιοσύνη. Όταν υποβάλλουμε τα αποδεκτικά στοιχεία αυτά για την εμπλοκή του Υπουργείου Δικαιοσύνης ξεκίνησαν δίκη κατά εμού. Με κατηγορία ότι συκοφαντώ την αστυνομία. Και φυσικά έρχονται όλοι να μου πούν ότι είσαι χαζή, γιατί το επόμενο θύμα του τράφικινγκ θα είναι η κόρη σου. Γι' αυτό λοιπόν την πήγαμε στην Ολλανδία το 2009, αλλά συνεχίσαμε τη δουλειά που κάναμε. Το 2011, μια ομάδα πολιτών ήρθε στο γραφείο μας και μας είπε ότι τους κατεδάφιζαν τα σπίτια, τα συνταγματικά δικαιώματα του κόσμου στη χώρα μας ανύπαρκτα. Το 2011 ξεκινήσαμε έρευνες και πάνω από 60.000 κατοικίες στον Πακού είχαν κατεδαφιστεί παράνομα για να φτιάξουν ένα πάρκο όπως είχαν αποφασίσει. Τον Αύγουστο του 2011 έδωσα μια συνέντευξη η οποία και δημοσιεύτηκε για την παραβίαση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στο Αζερβαϊτζάν. Δημοσιεύτηκε λοιπόν αυτή η συνέντευξη και μετά μας καταδάφησαν το δικό μας το σπίτι, το οποίο ήταν και τα γραφεία του Ιδρύματός μας τότε. Και χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση. Όλα καταστράφηκαν, βιβλιοθήκες, αρχεία, όλα. Και ε, υποτίθεται ότι υπήρξε μια απόφαση να μας αποζημιώσουν, τίποτα δεν πήραμε. Όλοι οι πολίτες λοιπόν στο Ζερμπαϊτζάν είναι αδύνατοι, ανίκανοι να προστατεύσουν τα παιδιά τους, την οικογένειά τους, το σπίτι τους. Και η βία φυσικά εξωθέσε βία. 20% του, της χώρας, 80% ε, μάλλον της χώρας είναι το τσιφλίκι των πολιτικών μας. Και τη χώρα την έχουν διαρρεμένη μεταξύ τους, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα τους οι υπουργοί. Οι συνάδελφοί σα επίση ε, είπαν ε, χτες ότι έχουμε πετύχει κάποια πρόοδο και ότι το Αζερβαϊτζάν κάπω θα βελτιωθεί. Και τώρα θα μπορέσουν να απελευθερωθούν πιο πολύ πολιτικοί κρατούμενοι κλπ. Όμως, σας ευχαριστούμε για το θέμα της ε, απλεθέρωσης, αλλά τι να το κάνουμε που βάζουν άλλους στη φυλακή. Τώρα έχω 148 άτομα στον κατάλογο πολιτικών κρατουμένων στην λίστα μου αυτή. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε. Τι προτείνουμε να κάνουμε σε τέτοιες καταστάσεις θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνονται πραγματικές πληροφορίες για το πώς έχει η κατάσταση στις χώρες μας. Φυσικά, η Human Rights Watch, η Amnesty International δίνουν πληροφορίες για τα θύματα κατασταλτικών μέτρων. Αλλά χρειάζεται πιο πολύ προσοχή για τους ακτιβιστές. Έχουμε πάρα πολλούς φιλήσυχους πολίτες στις φυλακές και έχουν φυλακιστεί μόνο επειδή έχουν α, επικρίνει, έχουν ασκήσει κριτική στον πρόεδρο. Στο μουσουλμανικό Αζερμπαϊτζάν προβάλλεται ως ε, σωτήρες της ε, περιοχής προστάτης από την Ισλαμική τρομοκρατία. Και η κατάσταση είναι ακριβώς ε, αντίθετη, γιατί ο Ιλχάμ Αλίεφ βασανίζει και φυλακίζει χιλιάδες ε, πολίτες και αυτός εξωθεί στην ρίζοσπαστικοποίηση. Και αυτό λαμβάνει χώρα στη χώρα μου όπως την ώρα που μιλάμε. Ο σύζυγός μου έχει δημοσιεύσει ακτοβιβλία για το Ισλάμ και για, τις, ε, για τους κινδύνους της καταστολής στον Κάφκασο. Και θυμάμαι πολύ καλύτερα μετά την ε, κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, όταν μιλήσαμε για την φρικτή κατάσταση του Ζερμπαϊτζάν. Οι εμπειρογνώμονες από την Ευρώπη μου είπαν ότι χρειαζόμαστε μια μεταβατική περίοδο. Και έδωσαν ως παράδειγμα την Αίγυπτο, τον Μουμπάρακ, τον Ασάντ, την Συρία. βελτιώνουν ε, βήμα προ βήμα την κατάσταση προ τη δημοκρατία και το Αζερβαϊτζάν υποτίθεται θα κινούνται προ την ίδια κατεύθυνση. Σήμερα λοιπόν. Τι έχει γίνει με τον Άσαντ. Δεν θέλω αύριο το Αζερβαϊτζάν να καταστεί Νέα Να θυμάστε ότι η επόμενη τέτοια κρίση θα είναι σε μια πρώην Σοβιετική μουσουλμανική χώρα το Αζερβαϊτζάν, το Κυριγιστάν. Ποιο ήταν ο Καμικάζη στην ε, Κωνσταντινούπολη τον Ιούνιο, στην Τσένη, Κυργιζή και Ουσμπέκη. Η βία εξωθεί σε βία και τέτοιοι δικτάτορες όπως ο Λιχάμα Λίγεφ δεν δίνουν καμία δυνατότητα για να βελτιωθούν τα πράγματα ειρηνικά στην κοινωνία των πολιτών, για να αλλάξει το καθεστώ τη εξουσία, ειρηνικά. Και τώρα η Ευρώπη αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα με πολλού ε, πρόσφυγε από τι Αραβικέ χώρε. Αν δεν υπάρξει αντίδραση και δεν υπάρξει δυνατότητα για μια ειρηνική μετάβαση στο Αζερμπαϊτζάν και στι άλλε πρώην σοβιετικέ ε, χώρες, οι πρόσφυγε θα είναι από τι δικέ μα χώρε στο μέλλον. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ τον χρόνο σα για την υποστήριξή σα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρώπη να υποστηρίξει τους πολιτικούς κρατούμενους, όλους τους. Να μην υπάρξει διάκριση βάσει θρησκείας. Εβραίοι, ε, χριστιανοί, μουσουλμάνοι, όλοι από κοινού, όλοι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στους καταλόγους μας για τους πολιτικούς κρατούμενους, για το Καραμπάκ τώρα. Γιατί δεν πετύχαμε την ειρήνη εκεί. Φυσικά παίζει μεγάλο ρόλο η Ρωσία. σε ό,τι αφορά τα όπλα στην Αρμενία, τα όπλα στο Αζερβαϊτζάν. Γιατί κάθε δικτατορός χρειάζεται έναν ξένο εχθρό. Έναν ξένο και έναν ε, εσωτερικό εχθρό. Πριν από την ψηφοφορία τον Απρίλιο, ο κόσμος ε, στο Αζερβαϊτζάν τι ζητήσε, ειρηνή, όχι, τρόφιμα ζητούσε. Αλλά Μετά άρχισαν τα σλόγγαν. Να, συνεχιστούμε το, να συνεχίσει ο πόλεμος, να ξαναπάρουμε το Καραμπάχ. Όλη η κοινότητα ζήτησε τον εκδημοκρατισμό, την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Στις τέσσερις ημέρες όμως αυτές, τον πόλεμο των τεσσάρων ημερών, ζητήθηκε και η χειρία. Ποιος ε, κέρδισε, ο Ιλχάμ Κέρδισε τον πόλεμο αυτό. Το 2004 δημιουργήσαμε στο Αζερβαϊτζάν το πρώτο και μοναδικό ανιαίο website ε, μεταξύ ε, Αζερβαϊτζάν και Αρμενίας. Αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία για την εξαγωγή διαλόγου Ξέρετε πώς μεγάλα είναι η καινούργια γενιά στη χώρα μας. Στην Αρμενία τους λένε ότι οι Τούρκοι και οι το Αζερμπαϊτζάν είναι οι τους. Αναλύουμε λοιπόν τα βιβλία της ιστορίας για να δούμε ποιοι ήταν ε, οι οι υπεύθυνοι για όλα τα δεινά του 19ου αιώνα. Οι Αρμένοι λέμε ότι είναι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται λοιπόν. Αυτά στα σχολικά βιβλία. Και όσοι επιδιώκουν ειρηνικέ λύσει, ε, του βάζουν φυλακή. Του λένε ότι είναι κατάσκοποι. Αρμένοι. Θα πρέπει λοιπόν να ενώσουμε τι δυνάμει μα. Οι δημοσιογράφοι, οι ακτιβιστέ, οι ευρωβουλευτέ, οι μουσουλμάνοι οι χριστιανοί οι Εβραίοι για να καταπολεμήσουμε τον εποτισμό και την δικτατορία, να ταχθούμε υπέρ τη ειρήνη και τη δημοκρατία για τη δική μα και τη δική σα ελευθερία. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάννου. Κύριε Γιάννου, την κόρη σα. Σα ευχαριστώ για αυτά που μα είπατε. Οπωσδήποτε θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το Αζερβαϊτζάν για να επιτύχουμε κάποια λογικά πράγματα και τα θέματα που αναφέρετε. τις συγκρούσεις με την Αρμενία νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει έναν ισχυρό ρόλο γιατί δεν ωφελεί κανέναν η κατάσταση ούτε την Αρμενία ούτε το Αζερβαϊτζάν Πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένα συμβιβασμό για τους ανθρώπους στην περιοχή. Και εγώ κατάχομαι από μια χώρα που είχε χωριστεί στα δύο. Ξέρω από την οικογένειά μου το τι σημαίνει πρακτικά για τις οικογένειε. Και με τον πόλεμο των τεσσάρων ημερών έχουν δει πως αυτοί που βάλαν την φωτιά ε, μετά κάναν τους πυροσβέστες. για να αναφερθώ στο ρόλο της Ρωσίας. Να είστε σίγουροι λοιπόν πως εδώ πάντα είναι ανοιχτέ πόρτες για σας. Και για σας συγκεκριμένα τώρα βέβαια που είστε κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα να ευχαριστήσω τις Ολλανδικές Αρχές που σας έδωσαν τόσο γρήγορα και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες άσυλο. Δεν σημαίνει αυτό έτσι εύκολα παντού. Και εύχομαι καλή επιτυχία στο μέλλον και να επιστρέψετε στη χώρα σας σε μια καλύτερη κατάσταση υπό καλύτερες συνθήκες. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.